Καλημέρα συνάδελφοι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση γιατί ο Επίτροπος Τίμεμαντς ε, χρειάστηκε να ασχοληθεί με ορισμένα πήγοντα θέματα πριν έρθει. Και πρέπει να φύγει και σύντομα χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση. Θα ξεκινήσω τη συνεδρίαση από πλευρά της Επιτροπής Ανάπτυξης. Χαίρομαι που είναι εδώ η κυρία Βαλεάνα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με τους ε, δύο επισκέπτες μας, Τίμερμαντς και Τζέφρι Σάξ και θα συζητήσουμε και την έκθεση πρωτοβουλίας για την εφαρμογή των ε, βιώσιμων στόχων. Έχω κάποιες ανακοινώσεις για την ΤΕΒΕ, αλλά, αλλά θα τις ε, κάνουμε στις 12 και 10 όταν θα λήξει η κοινή συνεδρία. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Βαλιάνα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που και πάλι ε, συνεδριάζουμε μαζί για ένα τόσο σημαντικό θέμα που είναι η βιώσιμη στόχη ανάπτυξης και το θεματολόγιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση όπως υπόθηκε έχουμε διάφορα θέματα, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο σκέψεων για μια βιώσιμη Ευρώπη με το 2030, το έγγραφο ε, σκέψεων και έχουμε καλέσει τον Επίτροπο Τίμερμανς που θα μας παρουσιάσει το θέμα και κατόπιν οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να υποβάλουν ερωτήσεις, αλλά πολύ σύντομα παρακαλώ, γιατί όπως υπόθηκε ο Αντιπρόεδρος ε, πρέπει να φύγει. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Τίμερμαντς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, συγγνώμη πρώτα απ' όλα που καθυστέρησα. Ε, το συχαίνομαι να καθυστερώ, αλλά ήταν ε, κάτι που δεν μπορούσα να αποφύγω. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Δεν θα αναφερθώ στην ιστορία των βιώσιμων στόχων ανάπτυξη, πώ προέκυψαν και τι ρόλο έπαιξε η Ευρώπη σε αυτό. Επιμένω όμω ότι ένα χρόνο μετά τον καθορισμό των ε, στόχων αυτών στα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υιοθέτησε μία προσέγγιση με δύο φάσει. Πρώτα απ' όλα θα περιέχονταν ω κύριο στοιχείο σε όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παράλληλα θα ξεκινούσαμε μία ε, θεωρητική αναζήτηση για να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την πολιτική μα αυτή για τις διάφορες ε, κλαδικέ πολιτικέ μετά το 2020. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το έγγραφο με τι σκέψει μα που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι το δεύτερο βήμα κοιτάζει την κατάσταση, πώς είμαστε δηλαδή, πού είμαστε τώρα και διαμορφώθηκε μετά από μια διαδικασία που τους περιέλαβε όλους. Ε, έμαθα πολλά από αυτήν την ε, ανταλλαγή απόψεων με πολλούς και νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε για τη διαμόρφωση των ε, πολιτικών μας στο μέλλον. Συζητήσαμε και εντός των υπηρεσιών μας, αλλά επίσης δημιουργήσαμε και μια πλατφόρμα υψηλού επίπεδου όπου συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του κειμένου αυτού και η διαδικασία αυτή της πλατφόρμας υψηλού επίπεδου με ενέπνευσε γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι συναντήθηκαν από αυτούς που ασχολούνται με την προστασία των ε, πτηνών μέχρι τις ε, επαγγελματικές ενώσεις ε, των εργοδοτών και καταλήξαμε σε συμφωνία για τις καθημερινές γραμμές. Και νομίζω ήταν πολύ θαραλέο. Και όλοι αυτοί ήταν πολύ θαραλέοι, έθεσαν τα θέματά τους, τα συνδικάτα, τα εμπορικά επιμελητήρια, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, άλλοι ενδιαφερόμενοι φορεί και κατάφεραν να καταλήξουν σε συμβασμού. Αυτό είναι ο τρόπο για να αλλάξουμε τον, τρόπο πιο βιώσιμο, τον κόσμο συγγνώμη, με, το, με πιο βιώσιμο τρόπο. Η κοινωνία νομίζω ότι είναι έτοιμη γι' αυτό. Έτσι είδα Ακόμη και ο επιχειρηματικό κόσμος ε, είναι πιο προετοιμασμένο από ότι η πολιτική. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να προωθηθεί αυτό το θέμα. Ο, ο κύριος μας στόχος θα είναι να έχουμε μια συνολική εικόνα και να θέσουμε την μελλοντική μας συζήτηση σε ένα ανώτερο επίπεδο αξιοποιώντας όσο περισσότερο γίνεται τις ε, επιστημονικές γνώσεις. Γιατί νομίζω ότι τα στοιχεία είναι αδιαφυσβήτητα αν και πολλοί συνεχίζουν να τα αμφισβητούν, αλλά είναι αδιαμφισβήτητα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το τονίσουμε και γραπτό. και πρέπει να μην υπάρχουν αυτές οι παρανοήσει που ε, υπάρχουν ακόμη στην κοινωνία ότι και αν δεν κάνεις τίποτα δεν θα αλλάξει τίποτα. Πρέπει να δράσουμε, να αποφύγουμε περαιτέρω επιδείνωση για να αποφύγουμε πολέμους και εμφυλίους πολέμους για αγαθά πρώτης ανάγκης όπως καθαρός αέρας ή πόσιμο νερό. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πραγματική αλλαγή και είμαστε σε καλή φάση για να το κάνουμε και το έγγραφο αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε τίποτα για το οποίο πρέπει να τρεπόμαστε αν συγκρίνουμε την ε, κατάσταση της ε, περιοχής μας με άλλες περιοχές του κόσμου. Αλλά όσο πιο γρήγορα και όσο πιο αποτελεσματικά κάνουμε αυτές τις αλλαγές τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα ωφέλη και μπορούμε να ηγηθούμε τι προσπάθειε ο κόσμο μα να καταλήξει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Το έγγραφο, νομίζω, επίση δείχνει ότι βεβαίω η προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι κάτι το οποίο θα μα κλείσει το σπίτι μα και θα μα κάνει να μην έχουμε τίποτα να χαρούμε. Όχι. Πρέπει να έχουμε μια συνολική λοιπόν προσέγγιση και όραμα. Αν δεν έχει κανεί, για παράδειγμα, κοινωνική βιωσιμότητα, δεν θα μπορέσει να πείσει ε, τι δημοκρατικέ κοινωνίε να αναλάβουν του κινδύνου για να γίνουν οι αλλαγέ που χρειαζόμαστε και να αξιοποιήσουμε και τι ευκαιρίε που αυτή η αλλαγή θα προκαλέσει. Ιδιαίτερα πρέπει να αποδείξουμε και να το δείξουμε σε όλου ότι ε, μπορεί να γίνει εάν ο καθένα παίξει το ρόλο του και να λάβει τι ευθύνε του. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι μόνο κάποιοι θα πληρώσουν, δεν θα το δεχτούν. Αλλά εάν δείξουμε ότι όλα τα τμήματα των κοινωνιών θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα φέρουν το βάρος που τους αναλογεί, τότε θα το δεχθούν. Νομίζω ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία, για παράδειγμα, της εκπαίδευσης όλα αυτά. Όχι μόνο να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία μας να καταλάβει τι σημαίνει βιωσιμότητα, αλλά να δημιουργήσουμε και μορφές εκπαίδευση που θα επιτρέπουν στην κοινωνία μας να προσαρμόζεται συνεχώ στι προκλήσει τη βιωσιμότητα. Πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνία μα στο γεγονό ότι η εκπαίδευση δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει όταν πάρει κάποιο πτυχίο. Είναι κάτι που πρέπει να κάνει σε όλη τη διάρκεια τη ζωή σου. Επίση, οι επενδύσει, οι ιδιωτικέ επενδύσει θα χρειαστούν. Πρέπει να καταργηθούν όλες οι ε, χρηματοπιστωτικές ε, διαδικασίες που πάνε αντίθετα στη βιωσιμότητα. Πρέπει να αλλάξουμε την οικονομία μα προ μια κυκλική οικονομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τα πρώτα βήματα προ αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε τρία σενάρια τα οποία αναφέρουμε. Ένα σενάριο μια συνολική λύση, ένα σενάριο που εν μέρη αντιμετωπίζει τι προκλήσει και ένα σενάριο που λέει Α τα κάνουν άλλοι, εμεί δεν ασχολούμαστε. Νομίζω ότι από τον τρόπο που τα ανέφερα καταλαβαίνετε τι προτιμώ. Αλλά τα κράτη-μέλη και άλλοι εμπλεκόμενοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσουν τελικά ποιο σενάριο θα προτιμήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Συνάδελφοι, ο καθένας έχει από ένα λεπτό για ερωτήσεις που θα θέλετε να θέσετε προς τον κύριο Αντιπρόεδρο. Ο Τζον Λάινεν, πρώτος. Ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγή, κύριε Αντιπρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι την επιτυχία. Πώς την μετράτε για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΑΕΠ δεν είναι πλέον η ενδεδειγμένη παράμετρος. Ποια κριτήρια χρησιμοποιούμε, έχουμε, θα τα αναπτύξουμε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, είσαστε υποψήφιος για τη θέση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουμε να πάρει τη θέση. Πώ θα αναδιοργανώσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσετε να συντονίσετε αυτό τι προσπάθειε για την επίτευξη του τεράστιου στόχου, διότι χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, χρειάζεται συντονισμό, χρειάζεται συνεκτική προσέγγιση. Αυτέ είναι οι δύο ερωτήσει που έχω για εσά. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λίτ. Ευχαριστώ, Φραντ. Πολύ ωραία αυτή η εισαγωγή. Ήμασταν μαζί σα στη Νέα Υόρκη με την Τάμα και άλλου από την Επιτροπή όταν ξεκίνησε το 2015. Άρα θέλουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά αυτού του στόχους τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχω δύο ρωτήσεις. Ένα στόχο είναι η κατανάλωση. Λοιπόν, εφοδιασμό, η κυκλιακή οικονομία, σημαντικό παράγοντα. Αναφερθήκατε στι επιχειρήσει. Θέλουμε, βλέπουμε μεταμόρφωση στην κλωστιφαντουργική ε, βιομηχανία, κάποιες αλλαγές πρόοδο σε κάτι μέλη. Έχουμε ευκαιρία εκεί. Έχουμε τις κατευθείας γραμμές ε, για τον ΟΣΑΙ, τη σωστή συμπεριφορά όσον αφορά για τα υποδήματα, τα κλωστοϊφοντηρικά, τα δερμάτινα. Είναι καλή ευκαιρία αυτή για τις επιχειρήσεις, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και να, κάνουν, να θέσουν οι επιχειρήσεις πρότυπα και να έχουμε και νομικά δεσμευτικούς κανόνες. Κάτι που ζητούμε εμείς για ορθή διαχείριση. Η Φιλανδία καταβάλει προσπάθεια και η γερμανική ε, κυβέρνηση προσπαθεί να το προωθήσει αυτό για την ε, σωστή προσέγγιση στο θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Αντιπρόεδρε. Έχω ερώτηση για την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Είπατε ότι το έγγραφο για τους πολλαπλούς εμπλεκομένους ενδιαφερομένους επηρέασε πολύ το έγγραφο προβληματισμού. Στην παράγραφο που αναφέρεται στην υπεύθυνη συμπεριφορά επιχειρήσεων, τη σωστή συμπεριφορά των επιχειρήσεων, τα αποτέλεσματα είναι απογοητευτικά αναφέρεται η σωστή προσέγγιση ε, και με δεσμευτικό τρόπο, με δεσμευτικά μέτρα στον αφορά τους πολλαπλούς εμπλεχομένους και είπατε ότι ίσως θα δεχόσαστε αυτή την προσέγγιση αναφερόμενο σε διάφορους δείκτες. Τώρα φαίνεται να αναγνωρίζετε μόνο το περίπλοκο ή ελλειπές ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι ένα εμπόδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα, για να πετύχετε του στόχου, τι προσέγγιση θα ακολουθήσετε στην επόμενη θητή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. κυρία Χόιμπαχ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την ε, παρουσίασή σα. Έχω μια γενικότερη ερώτηση σχετικά με τα σενάρια τα οποία αναφέρατε. Ε, αναφέρονται λοιπόν διάφορα σενάρια για το μέλλον και διαπίστωσα ε, για μεγάλη μου χαρά ότι το πρώτο σενάριο θεωρείται αρκετά πιθανό. Πώς μπορούμε όμως πώς μπορείτε μάλλον εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρετε τη δυνατότητα για αυτά τα δύο σενάρια τα οποία κανονικά ε, φαίνονται ανέφικτα ως προς την πραγματοποίησή τους. Τι ε, βλέπουμε ότι όταν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν ε, τις, ε, δεν καταβάλουν τις ίδιες προσπάθειες δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το σενάριο 3 είναι ε, κάπως ε, άσχημο, δηλαδή να δούμε πρώτα τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Βλέπω λοιπόν ότι αντί να ηγείστε Αντί να ηγείται μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την επιτεύξη των στόχων, μένετε πίσω. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νόιζερ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη ερώτηση. Όλες οι επιτροπές μας έμαθαν πολλά τα τελευταία χρόνια. Οι βασικές καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές ήταν Επιτροπή Περιβέλλοντος και Ανάπτυξης. Τώρα γίνεται μάχη μεταξύ των επιτροπών. Όλες οι επιτροπές θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη όσον αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ποια είναι η άποψή σας? Μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σαν εκλεγμένος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θα κάνετε? Θα έχετε επίτροπο αρμόδιο αποκλειστικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ίσως επιτροπή να υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα έχει αποκλειστική ευθύνη του στόχου τη βιασμή ανάπτυξη. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερη. Είδα μια πολύ καλή πρωτοβουλία για την περιοχή Ασία Ειρηνικού. Αναφέρονται σε ένα σημείο συγκεκριμένο. Λένε όλοι αυτοί οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη είναι στο τοπικό επίπεδο. Να πλησιάσουν λοιπόν αυτοί οι στόχοι τη πόλη, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη ΜΚΟ. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα. Ο κ. Γκερέρο Σαλών, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ένας από τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε είναι να υπάρξει άνισο επίπεδο εφαρμογής των στόχων αυτών από τα διάφορα κράτη-μέλη και πολύ άνισο μάλιστα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποχρέωση να δημιουργήσει μια δυναμική αλληλοστήριξης για να εφαρμοστούν αυτοί οι στόχοι. Έχετε πείρα εδώ και πέντε χρόνια ως αντιπρόεδρος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υψηλή εμπειρία. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να σκεφτούμε, όπως είπε ο Γιώ Λάινεν, όχι μόνο την ε, δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και την φυσιολογία, όχι μόνο την ανατομία, αλλά και τη φυσιολογία, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν από κοινού οι υπηρεσίε στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάλεμπαχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτά που μας είπατε. Μας είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξεφορτωθούμε τις αντιπαραγω... τα αντιπαραγωγικά κίνητρα παραγωγής. Χρειάζεται να δώσουμε λοιπόν ε, γρήγορα ένα μήνυμα για το ε, ποιε είναι οι προτάσει που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε του ε, αναπτυξιακού στόχου τη χιλιετία. Όχι μόνο σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και εμεί τι μπορούμε να κάνουμε, οι επιμέρου επιτροπέ. Χρειάζεται έγκαιρη πληροφόρηση έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φως σε κάποιες προτάσεις ή αν πρέπει να πούμε μισό λεπτό να δούμε πρώτα, να εξετάσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ είναι η τελευταία. Σύντομα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα συνεχίσω στα γερμανικά. Να συνεχίσω σε αυτά που είπε η κυρια μαισνερ ειναι τελευταια συντομα Κάντενμπαχ. Σήμερα λοιπόν έχετε εδώ τις ε, δύο επιτροπές για να συζητήσουμε τους ε, στόχου βιώσιμη ανάπτυξη που μα αφορούν όλους. Πρόσφατα είχαμε μια εκδήλωση για τους πράσινους ε, λιμένες. Και τα ίδια τα λιμάνια έχουν υποχρέωση να κάνουν ε, πράγματα έτσι ώστε να πετύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ίσως ε, είναι μια καλή λύση αυτό το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη, ίσως όχι. Όμως, εγώ θέλω να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και να τονώσουμε τους διάφορους κλάδους, διότι ακριβώ το θέμα αυτό αφορά όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Λίντα έχει το λόγο να τονίσω αυτό που είπαν και διάφοροι συνάδελφοι για την αλυσίδα ε, φωδιασμού και τη δέωση επιμέλεια αυτής της αλυσίδας. Αν δεν δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεχωριστά τα κράτη-μέλη θα αρχίσουν να θεσπίζουν δική του νομοθεσία. Το είδαμε αυτό με το κακάο, που η βιομηχανία λέγει ότι χρειαζόμαστε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοβουλία. Διότι έχουμε γαλλική προσέγγιση, γερμανική, το ίδιο στην κλωστοφοντουργία, όπω είπε η Αναλίζα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απομακρυνθεί από τη μανία με θελοντικέ προσεγγίσει που οι ίδιε οι επιχειρήσει ξέρουν ότι δεν έχει πετύχει. Και τέλο, για να θέσουν τι επιλογέ επιτάπητο. Σαν Βρετανοί, θεωρώ ανησυχητικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει επιλογέ που δεν είναι καλέ επιτάπητο. Η τρίτη επιλογή είναι σαν να, η επιλογή του να μην κάνουμε τίποτα. Και ο συντονισμό τη άλλη, τα διάφορα στάδια. Αν θέλετε τα κράτη-μέλη να το ενστερνιστούν, πρέπει να τα υποχρεώσουμε να συμμετάσχουν. Ε, και θα πρέπει να έχουμε και εξέταση από μοτίμους, να γίνεται σύγκριση, αντιπαράθεση μεταξύ χωρών. Πρέπει να κάνετε περισσότερα. Ανησυχώ όμω. Έτσι που αναφέρεται το ενδεχόμενο το 2, μπορεί να οδηγήσει τις χώρες να χρησιμοποιήσουν το τρίτο ενδεχόμενο. Πώς θα καθοδηγήσετε τη συζήτηση. Δεν θέλω να καταλήξουμε σε ένα από τα άλλα δύο σενάρια. Χρειάζεται κάποια ηγεσία στον αυτού του στόχου. Είδαμε στην Νέα Υόρκη ότι είπα εξετάζει όλη τη διαδικασία για του βιώσιμου στόχου. Θα πρέπει η Ευρώπη να υψώσει τον αίσθημά τη τώρα. Αν δεν το κάνουμε τώρα, ίσω όλοι αυτοί οι στόχοι ε, να εξαφανιστούν όπω και πολλέ άλλε πρωτοβουλίε στο ΙΕ μέχρι τώρα. Κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώ Λάινεν έκανε μια ερώτηση την οποία έκανα και, έκαναν και αρκετοί συνάδελφοι. Πώς λοιπόν μπορούμε να μετρήσουμε την επιτυχία. Νομίζω πως ε, σε κάποιο βαθμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ε, κάθε ένα στόχο βιώσιμης ανάπτυξης, να θέσουμε διάφορα ε, μέτρα αξιολόγησης και είπατε κι εσείς ότι χρειάζεται να σκεφτούμε νέους τρόπους μέτρησης της επιτυχίας και φυσικά να αναθεωρήσουμε όλο τον ε, ορισμό της επιτυχίας. Τι αποτελεί επιτυχημένο στόχο, ανάπτυξη ή κάτι άλλο. Ε, πρέπει να μετρήσουμε και το περιβαλλοντικό κόστος ε, στις αναλύσεις που θα κάνουμε. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα στοιχεία ποικιλοτρόπως. Και αυτό νομίζω θα φανεί και στο μέλλον ότι είναι αναγκαίο. Επίσης, αρκετοί από εσά με ρώτησαν πώς θα οργανώσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον γίνω πρόεδρος της μετά τις εκλογές και τι θα κάνω ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τους στόχου βιώσιμης ανάπτυξης. Θεωρώ τον εαυτό μου κύριο υπεύθυνο και αρμόδιο για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ακριβώς διότι ε, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν όλους τους ε, τομείς της ε, Κομισιόν. Και οι δραστηριότητε ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίση να αξιολογούνται με βάση του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρώ ότι όλοι οι τομείς δραστηριότητας ε, της Κομισιόν μπορούν να συνδεθούν με έναν ή περισσότερους από τους 17 στόχους ε, αυτούς. Και νομίζω πως θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς για τη γενικότερη λειτουργία της Κομισιόν. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος ε, αρμόδιος και υπεύθυνο ε, θα πρέπει να είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψει και να οριοθετήσει τις δραστηριότητές της ε, ως προς την επίτευξη των στόχων. Τώρα, η αλυσίδα εφοδιασμού. Συμφωνώ μαζί σας. Ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά. Χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στην κλωστοϊφαντουργία διότι ακόμα και οι πιο προηγμένοι ε, τομείς της κλωσοφαντουργίας δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Δεν μπορούν να μας πούν αν το βαμβάκι θα είναι βιώσιμο ως ε, ύλη στο μέλλον. Δεν ε, γνωρίζουν ή δεν μπορούν να γνωρίζουν αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις σχετικά με την εργασία, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Ε, είμαστε πολύ κοντά στους στόχους του ΩΣΑ, όμως νομίζω πως ε, θα έπρεπε να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι. Μετά, ε, να πω ότι σίγουρα η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και την κοινωνία και την δημόσια υγεία. Πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν πλέον μικροπλαστικά στα, στην, στα υφάσματα. Υπάρχουν Συγκεκριμένε προτάσει και όχι περισσότερες, ακριβώς διότι η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λύγει σύντομα και θα είναι έργο της επόμενης Κομισιόν να συμπληρώσει με νέους ε, στόχους, με νέες προτάσει. Φυσικά επήγει το θέμα. Ε, αν ήταν στο χέρι μου θα ξεκινούσαμε ήδη δουλειά και νομίζω πως έχουμε πολλά να κάνουμε, διότι ξέρετε πως ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε και πρόβλημα ως προς την στρατολόγηση νέου ταλέντου, διότι η γενιά της ε, χιλιετίας έχει αλλάξει νοτροπία. Έχουμε λοιπόν το χρόνο με το μέρος μας, έχουμε και τους πολίτες με το μέρος μας. Τώρα, γιατί τρία σενάρια. Σήμερα άκουσα τις ίδιες επικρίσεις ε, με πριν από δύο χρόνια, όταν είχαμε παρουσιάσει πέντε σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης. Δηλαδή, ρωτηθήκαμε και πάλι γιατί έχουν συμπεριληφθεί σενάρια ανεπιθύμητα. Διότι αυτά συζητιούνται και στα κράτη-μέλη. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και να δείχνουν ε, το τι θέλουν. Ας τα αφήσουμε λοιπόν να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Διότι είτε το θέλουμε είτε όχι και τα τρία σενάρια εκτός από τη δημόσια διαβούλευση με τα κράτη-μέλη είναι ε, σενάρια που θα αφήσουν να διαφανεί η θέση των κρατών μελών. Επίσης, νομίζω πως ε, δεν είναι σημαντικό μόνο το πώς θα οργανωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πώς θα εργαστεί. Και η Task Force, αυτή η πλατφόρμα, είναι κάτι που θα ήθελα να συνεχιστεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναπτύξουμε τις ε, λεπτομέρειες και αυτή η πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς είναι κάτι το οποίο ε, θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι ειδικά για περιβαλλοντικά ζητήματα δεν θα είχαμε καταφέρει να ε, δημιουργήσουμε μία τόσο ε, καλή μελλοντοστραφή στρατηγική αν δεν είχαμε την ε, συμμετοχή όλων. Τέλος. Με ρωτήσατε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις ε, θα γίνουν εκεί που πρέπει, ότι θα αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα κτλ. Νομίζω πως αυτό θα γίνει μέσω των κατάλληλων εργαλείων και εμείς είμαστε εκείνοι που θα πρέπει να παρέχουμε αυτά τα εργαλεία. Μπορούμε να δείξουμε μεγάλη φιλοδοξία ή και να θεσπίσουμε ένα αυστηρό πλαίσιο αρκεί να υπάρχει ε, μακροπρόθεσμος ορίζοντας και να μην αλλάζουμε άποψη και πορεία κάθε λίγα χρόνια. Νομίζω πως ε, αν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο τότε οι επιχειρήσει θα προσαρμοστούν σε αυτό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Οι δύο επιτροπέ μα θα υθετήσουν κοινή έκθεση στρατηγική που θα τροφοδοτήσει συζήτηση πριν από τη Σύνοδο του CBU και θα ενημερωθεί και το βήμα συζητήσεων υψηλού επίπεδου για το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Καλή τύχη για την πρόθεση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης κατά το υπόλοιπο της θητείας. Εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα δώσω το, την προεδρία στη Λίντα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Αρχίσαμε καθυστερημένα αλλά καταφέραμε να προχωρήσουμε αποτελεσματικά και να υποβάλουμε αναλυτικές ερωτήσεις. Στο επόμενο σημείο θα είναι μια παρουσίαση μιας μελέτης που ανατέθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης και αφορά την προσέγγιση της Ευρώπης όταν αφορά την εφαρμογή, την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, βέλτιστες πρακτικές και το μέλλον. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε ε, ε, έχουμε τη Eurostat παράγει στατιστικά στοιχεία αλλά δεν κάνει σύγκριση κατάλληλη. Θέλαμε ενδελεχέστερη ανάλυση για να δούμε πώ θα πάει η Ευρώπη στον αφορά του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό κάνει η μελέτη. Έχουμε δύο εμπειρογνώμονε εδώ σήμερα, την Ingeborg Nischoy και η Elizabeth Χέγκε. Η κυρία Nischoy είναι από τη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, εμπειρογνώμονα που τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, που ξέρει θέμα θέματα, και Elizabeth Χέγκε που είναι ερευνήτρια του Ινστιτούτου Βιώσιμη Ανάπτυξη και, και αναλύει και τι διεθνεί σχέσει. Θα σας δώσουμε λοιπόν το λόγο για να κάνετε μια παρουσίαση. Να κάνετε την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω στη δεύτερη διαφάνεια. Ήλπιζα ότι θα παρέμενε ο κ. Τιμερμάν και να του δείξω τη διαφάνεια. Αυτό ήθελα, αλλά δυστυχώ ε, δεν είναι εδώ. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που δίνετε για την, μέσω τη ανάθεση τη μελέτη, να κάνουμε μια γενικότερη επισκόπηση τη διακυβέρνηση την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξη και τα πρώτα μηνύματα ήδη έχουν διαφανεί ε, ότι είναι θετικά. Ελπίζουμε ότι αυτή η μελέτη δεν θα είναι ε, μια μοναδική μελέτη, αλλά θέλουμε να αποτελέσει μια βάση για το Κοινοβούλιο, ώστε όλοι να το χρησιμοποιήσουν το έγγραφο σαν εγχειρίδιο. Έχει ένα μεγάλο παράρτημα που αναλύει όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει συνεργασία, συνεργασία για δράση, να προωθήσουμε τους στόχους Και έτσι χάρη, ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους ε, για τη βοήθεια. Ευχαριστώ επίσης και τη Γραμματεία του Ευρωκοινοβουλίου. Η μελέτη ξεκίνησε όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα είχε παραλύσει, ε, είχε πετρώσει, δεν εκινεί το καθόλου. Τελειώσαμε τα Χριστούγεννα λοιπόν. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ανάλυση αντίδραση στο έγγραφο προβληματισμού. Τελικά κάτι έγινε, προχωρήσαμε και υπάρχουν κάποια σχόλια. Συχνά χρησιμοποιώ αυτή τη διαφάνεια και αυτές τις αναφορές. Η πρώτη φράση αναφέρεται στην, καθολική, στην καθολικότητα, την αρχή της καθολικότητας. Και το, η δεύτερη φράση αναφέρεται στη διακυβέρνηση. Εκεί εστιαστήκαμε. Δεν είναι ένα στο αποτέλεσμα, αλλά γενικότερα στην διακυβέρνηση, στην προσέγγιση. Και αυτό που ανέφεραν και ερωτήσει. Τι γίνεται με το συντονισμό, με τις γενικές αρχές. Να μπούμε στο στοιχείο της καθολικότητας, που αφορά την επιχειρηματολογία. Γραφική παράσταση για τους δείκτες της ανάπτυξης αναχώρα έχουν ξεχωριστέ αφετηρίες οι χώρες, αλλά όλε πρέπει να κινηθούν προς την βιωσιμότητα, προς την περιοχή της βιωσιμότητα. Είναι, πρέπει το ίχνος μας να μειωθεί. Ε, το GSR έχει παράγει μια ανάλογη γραφική παράσταση, σας δείξουμε. Παρακάτω. Βλέπουμε το στοιχείο της καθολικότητας από εθνική έποψη. Κάθε χώρα, κάθε φορέας πρέπει στο εσωτερικό να εξετάζει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, να εξετάζει και την εξωτερική πτυχή και πώς διασυνδέονται οι εσωτερικοί με την εξωτερική πτυχή και ποια είναι η ελληλεπίδραση. Όλα πρέπει να εξετάζονται με το φακό της βιωσιμότητας. Και ήδη στο σενάριο με βάση όλα αυτά βλέπουμε ότι το σενάριο 3 δεν ταιριάζει με το θεματολόγιο και τους στόχους του 2030. Έχουμε εδώ το σύστημα συντεταγμένων και τους στόχους. Καλύπτουμε και τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 και πέρα. Και εστιαζόμεθα στο τι γίνεται σε επίπεδο κοινοβουλίων. Αυτή είναι η αξία για τις χώρες, τις 28 χώρες. Όλες οι χώρες κινούνται εφαρμόζουσε στις βέλτιστες πρακτικές. Στην τελική ευθεία εξετάζουμε και χώρες οι οποίες δεν είχαν δραστηριοποιηθεί τόσο πολύ. Η Ελίζαμπεθ σε λίγο θα αναφέρει τα αποτελέσματα αναχώρα και φτάνουν στις συστάσεις προς το Κοινοβούλιο σχετικά με το ψήφισμα που είναι μια αντίδραση στο έγγραφο προβληματισμού. Εξετάσαμε αυτά τα 7 στοιχεία της διακυβέρνησης που αναφέρονται εδώ αριθμητικά. Συνοπτικά παρουσιάζω ότι τα ξέρετε. Το θέμα των πολλαπλών επίπεδων, του κατάλληλου συντονισμού των εξωπιπέδων, συντονισμού μεταξύ φορέων, μεταξύ τομέων. Βλέπετε τα επίπεδα, τους τομείς και τους φορείς στη γραφική παράσταση. Προσθέτουμε επίσης και τις γνώσεις που υπάρχουν, το θέμα της εποπτείας, πολιτική, εργαλεία, μακροπρόθεσμες προοπτικές. Ίγκα, είναι στη μελέτη σου όλα αυτά. Έχετε τη μελέτη, γιατί εγώ δεν βλέπω, δεν βλέπω από εδώ τις λεπτομέρειες που δείχνετε στα γραφήματα. Είναι δύσκολο να τα διακρίνουμε. Μπορείτε να πείτε σε ποιες σελίδες είναι, έχουν τη μελέτη, αν πείτε τις σελίδες να μπορούν να... Εδώ είναι στο παράρτημα. Άμα ανοίξετε το παράρτημα, είναι αυτοί οι πίνακες. Μελέτη είναι πίσω-πίσω. Δεν θέλω να κοιτάτε τη διαφάνεια, έτσι απεικονίζω, έτσι δίνω μια ιδέα για το όλο προϊόν. Page 163. 160, kind of the second half. Στο δεύτερο κομμάτι. Περάστε τη μέση και πηγαίνετε λίγο προς τα πίσω και θα τα βρείτε όλα αυτά. Α, τώρα τα μέλη που το έχουν διαβάσει ξέρουν. Λοιπόν, δεν έχετε αντίγραφα, το προσωπικό παρακαλώ να μοιράσει τα αντίγραφα του εντύπου, τόσο ώστε τα μέλη να έχουν μπροστά τους το έγγραφο. Αναλύσαμε λοιπόν όλες τις διαθέσιμες ε, μελέτες για τις χώρες που εφαρμόζονται εθελοντικά και υποβάλλονται αναφορές από τις χώρες εθελοντικά στον ΟΗΕ. 24 κράτη-μέλη έχουν συμμετάσχει. Είδαμε και τα δελτία για το δίκτυο των ευρωπαϊκών ε, βιωσιμότητας, ε, ο ΩΣΑ, τις διάφορες αναλύσεις. Προσεγγίσαμε σε αυτά ερωτήσεις. Είχαμε μια συνέντευξη ανακράτως μέλος και είδαμε ποιες είναι οι δραστηριότητες στα κοινοβούλια. Και εκεί κάναμε διάφορες συνεντεύξεις και επαφές. Καλή θα ήταν μια διεύρυνση προσέγγισης του προβληματισμού ανάλυση στο τι γίνεται σε επίπεδο κρατών μέλων και αυτό θα κάνει τώρα και η Ελίζα Ναι, κοιτάξτε. Στα δελτία των χωρών, τι κάναμε. Εξετάσαμε τα αυτά σημεία. Τα 7 ερωτήσει. Ποιο είναι το επίπεδο πολιτική προσπάθεια, στρατηγική, τι γίνεται με τον οριζόντιο συντονισμό, με τον κάθετο συντονισμό, συμμετοχή των ενδιαφερομένων, των εμπλεκομένων φορέων, παρακολούθηση, αναθεώρηση, ε, εργαλεία, αξιολόγηση, μακροπρόθεσμες προοπτικές, σχετικοί μηχανισμοί τα 7 σημεία. Έχουμε παράδειγμα, οι διαφάνειες είναι πολύ δυσανάγνωστες πράγματι. Βάζοντας όλες τις πληροφορίες λοιπόν στα δελτία των χωρών, κάναμε ομαδοποίηση ανάλογα με τις ερωτήσεις. Εδώ βλέπουμε την ερώτηση ποιο ηγείται, ποιο δικεί όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων των βιωσίμων, μέσω οποίων μηχανισμών, εάν υπάρχει οριζόντιο συντονισμό. Θα δείτε πιο ευανάγνωστου πίνακε στην έκθεση, στο κεφάλαιο 3. Μία από τι προστιθέμενε αξίε τη μελέτη είναι ότι δεν περιοριζόμαστε σε απλή περιγραφή τη διαδικασία υλοποίηση και του μηχανισμού διαχείριση τη χώρα, αλλά αναπτύσσουμε και μεθοδολογία αξιολογήσεω επιδόσεων χωρών μέσω των 7 αυτών θεμάτων. Για την ερώτηση 1 που βλέπουμε εδώ, που αφορά τη στρατηγική, το επίπεδο δέσμευση προσπάθεια στρατηγική, δώσαμε ένα βαθμό σε μια χώρα αν έχει διατομιακή στρατηγική, παρόλο που δεν έχει επικαιροποιηθεί πρόσφατα αυτό. Δύο βαθμού. Αν η στρατηγική το σχέδιο δράση δημιουργήθηκε πρόσφατα, επικαιροποιήθηκε με του στόχου διώσεων ανάπτυξη. Τρει βαθμού. Αν η στρατηγική η σχέδιο φαίνεται ότι είναι κάτι επιχειρησιακό, που σημαίνει ότι υπάρχουν σαφεί στόχοι, τρόποι προσμέτρηση και δράση. Και τέσσερι βαθμού. Αν η σχετίζεται με του εθνικού προπολογισμού. Εδώ βλέπετε μια συνόψιση της ε, αξιολόγησης που κάνουμε για κάθε χώρα με βάση τις 7 αυτές κατηγορίες. Εάν ε, έχει όλο το κεκάκι, σημαίνει ότι έχει, τέσσερα, έχει πάρει τέσσερις πόντους. Αν δεν έχει καθόλου κεκάκι, δεν έχει πάρει κανένα πόντο. Αυτά είναι στη σελίδα 91 της μελέτης. Οπότε οι περισσότερες χώρες έχουν ε, επικαιροποιήσει την ε, στρατηγική τους ή το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης που δεν το έχουν όλες οι χώρες. Ανάλογα λοιπόν με τη φύση του στρατηγικού χαρακτήρα της ένταξης ε, των στόχων της ανάπτυξης στην πολιτική τους και με βάση και την πολιτική βούληση οι στόχοι αυτοί είναι λιγότερο ή περισσότερο λειτουργικοί. Η περισσοτερο λειτουργικη η φιλανδια και η Δανία είναι οι πιο προηγμένες. Άλλες χώρες συνδέουν όλο και περισσότερο με τον προπολογισμό την στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη όπως η Σλοβενία. Επίσης, πολλές προσπάθειες έχουν γίνει και για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Οι περισσότερες χώρες έχουν κάνει πολλές προσπάθειες γι' αυτό, ορισμένες μάλιστα, σχεδιάζουν την στρατηγική τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνεργασία με αυτούς τους φορείς, όπως ε, το Λουξεμβούργο και την Γαλλία. Ορισμένες χώρες έχουν σαφείς μηχανισμούς συνεργασίας και συντονισμού των πολιτικών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ Υπουργείων και με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Πολλέ έχουν ε, ε, τακτικές εκθέσεις για το θέμα αυτό και επικαιροποιούν τους δείκτες τους και επίσης τι αναθεώρηση γίνεται. Η Φιλανδία και η Γερμανία κάνουν ε, αξιολογήσεις των ε, ε, προγραμμάτων τους από ανεξάρτητους ομοτήμους. Βλέπουμε πού σχεδιάζονται νέες δραστηριότητες, που δηλαδή υπάρχουν θέματα να εξελίξει. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Σλοβακία. Έγινε μια προσπάθεια να κάνουν προβλέψεις και είδαν έξι προκλήσεις μέχρι το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θέλουν να εντάξουν στην εθνική του στρατηγική με σαφείς στόχους, δείκτες και ακόμη πιο σημαντικό, θα συμπεριλάβουν τα θέματα αυτά στο σχέδιο επενδύσεών τους. Λοιπόν, συνοψίζοντας, πολλές δραστηριότητες βρήκαμε σε σχεδόν όλες τις χώρες. Δηλαδή, οι θεσμοί και οι υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή και αυτό ανεξάρτητα από τον πολιτικό προσανατολισμό των κυβερνήσεων. Αλλά βεβαίω πολλά μπορούν να γίνουν ακόμη. Ορισμένα μάλιστα είναι και εύκολα. Εύκολα θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Για παράδειγμα θα μπορούσαν ε, περισσότερε χώρε να έχουν ε, επιστημονικέ επιτροπέ για να παρακολουθούν την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξη. Και επίση θα μπορούσαν να ελέγχουν κάθε νέα πολιτική για να δουν αν περιλαμβάνει στόχους βιώσιμη ανάπτυξη και θα μπορούσαν επίσης να εντάξουν όλες ε, τις διαστάσεις βιώσιμης ανάπτυξης που δεν έχουν ακόμα εντάξει σε όλες τις πολιτικές. Επίσης, και αλλού υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης για πιο δύσκολα θέματα. Ο συνδυασμός της εσωτερικής με την εξωτερική διάσταση, ορισμένες χώρες δυσκολεύονται, δεν ξέρουν πώς ακριβώς να το επιτύχουν. Και επίσης, δεν καταφέρουν πολλές χώρες να συνδέσουν τους, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με τον προϋπολογισμό τους. Τώρα είναι, σύντομα παρακαλώ. Στη σελίδα 59 επίσης κάνουμε μια επισκόπηση των συμβάντων σε ενωσιακό επίπεδο. Στη σελίδα 60 συγκεκριμένα. Εδώ βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές ε, κολυσιεργεί και αναβάλει για αργότερα τις προσπάθειες αυτές. Ε, μετά βλέπετε τα 7 σημεία της ε, διακυβέρνησης, πώς ε, τα εφαρμόζει η Κομισιόν. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη εσωτερικού συντονισμού. Είναι πολύ καλή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να κάνει αυτό το συντονισμό και είναι πολύ καλή και η αντίστοιχη επιτροπή του Συμβουλίου. Αλλά πρέπει να κάνουν ακόμη περισσότερα. Και το βασικό μήνυμά μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα. Πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική δύο επιπέδων. Να δημιουργήσει μια επιτυχή δυναμική δύο επιπέδων. Όλα τα θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο. Πρέπει να εργαστείτε περισσότερο, να συνεργαστείτε περισσότερο με τα κράτη-μέλη. Η ομάδα εργασία του Συμβουλίου θα ήταν ένα καλό συνομιλητή. Και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα καλό μηχανισμό διακυβέρνηση για να γίνει μια συζήτηση, μια παρακολούθηση τη εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Θα έπρεπε να διευρυνθεί βέβαια το εξάμεινο για να γίνει αυτό. Αλλά έχει έννοια από πλευρά γενικά διακυβέρνηση. Για παράδειγμα και η επισκόπηση περιβαλλοντική ε, εφαρμογή είναι μία άλλη δυνατότητα συζήτηση για του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να συνεργαστείτε με τι εθνικέ κυβερνήσει. Να, εδώ βλέπετε. Σε πορτοκαλί είναι οι χώρε όπου τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ειδικέ προβλέψει για την εφαρμογή των στόχων του θεματολογίου 2030. Ξέρω ότι το έχετε συζητήσει αναλυτικά κι εσείς αυτό, πώς ακριβώς να προωθήσετε τους στόχους αυτούς. Δείτε τι κάνει η Δανία για παράδειγμα. Υπάρχει ένα δίκτυο και ένα σημείο εστίασης για τα θέματα αυτά. Ούτω ώστε όλες οι επιτροπές του Κοινοβουλίου να ασχολούνται με αυτά. Αυτό θα μπορούσε να σας εμπνεύσει. Πρέπει λοιπόν να μην περιχαρακώνει ο καθένας ε, την ε, ε, τομεακή του πολιτική για τα θέματα αυτά. Και γενικότερα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό που υπάρχει μέσω της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Θα μπορούσαν να υπάρχουν, για παράδειγμα, συναντήσεις ε, μεταξύ όλων των αρμόδιων επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συγκεκριμένε προτάσει κάνετε. Είναι πολύ περίπλοκα ορισμένα διαγράμματα, δεν μπορούσα να τα παρακολουθήσω, αλλά το βασικό μήνυμα είναι αυτό. Γιατί το Κοινοβούλιο τώρα σκέφτεται πώς να οργανώσει τη διακυβέρνηση της εφαρμογής των στόχων αυτών και είναι καλό να εξαγάγουμε διδάγματα. Είχαμε μια συνάντηση πριν από δύο χρόνια περίπου με τα Εθνικά Κοινοβούλια για το θέμα αυτό. Τότε όμως δεν υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά νομίζω ότι έκτοτε έχει βελτιωθεί η κατάσταση και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά. Οπότε, να περάσουμε στην επόμενη μελέτη. Έχουμε τον καθηγητή κύριο Βανίπεσελ, την Εύα Φούμαν, αλλά θα μας τα πει η κυρία Βαλιάν καλύτερα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προετοιμασίες για την έκθεση των ΟΕΕ Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε την κυρία Εύα Φούρμαν, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής της Φιλανδίας Τη Επιτροπή Ειδικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και είναι και διευθύντρια του Ινστιτούτου ΣΑΙΚΙ που είναι το Φιλανδικό Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μα δίνετε να σας παρουσιάσουμε την παγκόσμια προοπτική. Είμαι εδώ με τους ε, συναδέλφους μου και τον ε, καθηγητή κύριο Βαν Ήπερσέλε να ζητήσω συγγνώμη για ε, το ότι απουσιάζει ο κύριος ε, Μέσερλη, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτήν την μπάλα. Νομίζω πως αυτή, αυτή η μπάλα, αυτό το σχήμα αντιπροσωπεύει την ε, γη και το πως είμαστε όλοι συνδεδεμένοι και πως όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η λέξη κλειδί είναι με τα μεταβολές. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν μεταβολές σε έφτατο χρονικό διάστημα και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να κινητοποιηθεί τόσο η επιστήμη όσο και η απόκτηση γνώσης. Εκπροσωπούμε λοιπόν μια ομάδα 15 επιστημόνων και το 2016 μας ζητήθηκε να ε, συντάξουμε μια έκθεση για τα Ηνωμένα Έθνη. Έξι από εμάς ε, είμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 από εμάς ε, Ευρωπαίοι και νομίζω πως η ομάδα μας είναι αρκετά ενδεικτική ε, και ολοκληρωμένη. Σε τι εστιάζει λοιπόν η έρευνά μας, ε, στην διαπαφή της επιστημονικής πολιτικής και στην συμπερίληψη της επιστημονικής γνώσης στην πολιτική, αλλά και της επιστημονικής μεθοδολογίας και της ε, διεπιστημονικότητας. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε όλη την ε, γη με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες ε, περιοχές ή συγκεκριμένες χώρες. Είναι η πρώτη έκθεση που ζητήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, που ζητήθηκε από τις κυβερνήσεις. Η επόμενη έκθεση θα ξεκινήσει με την επόμενη τετραετή περίοδο, από το 2020 δηλαδή. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα θετικά. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, υπάρχουν και πολλά θετικά τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρωπότητα γενικότερα. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι πράσινες, έχει σημειωθεί, αρκετή πρόοδος ως προς αυτό, αλλά υπάρχουν και πολλές προκλήσεις. Υπάρχει ένα σημείο καμπής ως προς τα κοινωνικά ζητήματα και νομίζω πως αυτό δείχνει πως πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στα περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και στα κοινωνικά και ιδιαίτερα στις ανισότητες που παρατηρούνται εντός μιας χώρας. Παντού στον κόσμο υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, υπάρχει το ίδιο μοτίβο όπου το, τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας απομακρύνονται όλο ένα και περισσότερο από τα υπόλοιπα και οι ανισότητες λοιπόν αυξάνονται. Εντός μιας χώρας λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι μόνο η φτώχεια αλλά οι κοινωνικές και πολιτικές ανισότητες ως προς το περιβάλλον. Το σημείο καμπής εδώ είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά και θέματα πολυμορφίας. φαίνεται και στην έκθεση την, της Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να σας δείξω και ότι ε, η περιβαλλοντική διάσταση έχει άμεση σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη και την ικανότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει τους στόχους για αυτή. Υπάρχουν λοιπόν στην Ευρώπη τάσεις προς τα πίσω. Υπάρχει αυξανόμενη τάση εθνικισμού, λαϊκισμού. Βλέπουμε ομάδες οι οποίες πέφτουν σε πολλές παγίδες ακριβώς διότι το στόχος είναι ένα συγκεκριμένο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης και χάνουμε λοιπόν τους υπόλοιπους. Όλα αυτά θα τα διαβάσετε στην έκθεση. Τα επόμενα λοιπόν 10 χρόνια πρέπει να αλλάξουμε νοτροπία ως προς το ότι αποτελεί μια μεταβολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μεν ε, να εξετάζει το ζήτημα, όμως απομακρύνθηκε από κάποιους ε, στόχους εις βάρος κάποιων άλλων. Βλέπουμε ότι, η, ότι δόθηκε έμφαση στην οικονομία και έχει έρθει η ώρα λοιπόν να πάρουμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στους ε, τρεις ε, κύριους ε, στόχους, το περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία. Μπορούμε να τους συνδυάσουμε, αλλά και οφείλουμε να οριοθετήσουμε ε, το περιβαλλοντικό σκέλος ε, και το κοινωνικό από το οικονομικό. Και παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη γενικά τα πάμε καλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, χώρες όπως η Μπουρκίνα Φάσο και πολλές άλλες που απέχουν πάρα πολύ από τους στόχους αυτούς. Βέβαια υπάρχουν και τα λαμπρά παραδείγματα των βόρειων χωρών, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεν αυτή η πράσινη γραμμή και υπάρχουν τα θετικά, όμω κοιτάξτε και τι κόκκινε γραμμές και πόσε χώρε βρίσκονται κοντά σε αυτέ. Τώρα, στην έκθεση έχει γίνει μια μελέτη όπου προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα για να γίνει μια ανάλυση των ε, συνδέσεων Θέλουμε να, να δώσουμε έμφαση σε ε, συγκεκριμένα συστήματα και παρατηρούμε ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Παρά το γεγονός ότι είναι εύκολο να διαλέξουμε τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, που μας βολεύουν, υπάρχουν πάρα πολλοί ανεκπλήρωτοι. Υπάρχουν ωφέλη αλλά και μειονεκτήματα και χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στις ελλείψεις και να εντοπίσουμε τους ε, σημαντικούς τομείς, ε, τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης έτσι ώστε να τους βελτιώσουμε. Και κάτι άλλο που δεν φαίνεται στις ε, διαφάνειες που βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει στην ε, μελέτη, είναι ότι έχουν γίνει ελάχιστες έρευνες όσον αφορά τις ε, διασυνδέσεις ανάμεσα στους διάφορους τομείς πολιτικής και νομίζω πως θα ήταν πολύ καλό να εξεταστεί αυτό από τους ερευνητές. Βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, ότι οι κυριότερες προκλήσεις δεν ε, βρίσκονται στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιες ροές λοιπόν που είναι μη βιώσιμες, αφορούν όλο τον κόσμο και έχουν ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στις ε, δύο άκρες και στην πηγή αλλά και στον, στο τέλος της ροής αυτής. Μόλυνση, για παράδειγμα, του περιβάλλοντος, ρήπανση, ε, ακτική. Στην έκθεσή μας, ε, λοιπόν, δίνουμε έμφαση στο πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτήν την ε, αλλαγή. Η διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική. Η διακυβέρνηση όμως πρέπει να είναι παγκόσμια και ευρύτατη. Πρέπει να, να δούμε ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη και εννοώ τη συνεργασία τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και με το ευρύ κοινό. Μόνοι μας δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, ούτε, ένα, ούτε μια χώρα μόνη της μπορεί. Όπως είπε και ο πρόεδρος ε, Τίμερμανς, υπάρχει ε, μια τάση συνεργασίας και αυτό είναι κάτι το θετικό. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει πολιτική ηγεσία σε υψηλό επίπεδο έτσι ώστε να σημειωθεί η πρόοδος και όχι μόνο ε, σε μεμονωμένες πόλεις. Χρειάζεται η πρόοδος να είναι γενικότερη. Και τι μπορεί να κάνει ο καθένας ε, από εμά. Ε, οι αποφάσεις είναι μεν προσωπικές, όμως και εδώ πρέπει να υπάρχει διασύνδεση. Ως προς ε, το οικονομικό σκέλος τώρα, να πω μόνο ότι φυσικά πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος με τους πολίτες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σίγουρα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο. Ο διάλογος όμως είναι κέρια σημασία, διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι μεν σημαντική, αλλά δεν είναι μονόδρομος. Επίσης, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είναι εξίσου σημαντική. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά, να στηριχθεί η κυκλική οικονομία, για παράδειγμα, και εδώ βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει σημειώσει αρκετή και ικανοποιητική πρόοδο. Σε ό,τι αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία, θα πω μόνο ότι και εδώ πρέπει να αλλάξει το σύστημα Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να συνεργαστούμε με τις ε, τοπικές κοινότητες έτσι ώστε να κινητοποιηθούν τόσο οι πολίτες όσο και η έρευνα. Όμως, η επιστήμη έχει και πολλά και να Εστιάζει μόνο σε συγκεκριμένες προτεραιότητες και ε, χρειάζεται να στηρίξουμε τους ε, τομείς που έχει παραβλέψει η επιστήμη έτσι ώστε να βοηθήσουμε ε, και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο την επιστημονική πρόοδο. Στη δομή λοιπόν ε, της ε, πρότασης μας εξετάζουμε ορισμένα συγκεκριμένα συστήματα, ορισμένα συγκεκριμένες μεθόδους, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βλέπουμε ότι η διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική, βλέπουμε ότι αναλύουμε την οικονομία, την ε, συμπεριφορά και τον τρόπο που γίνεται αυτή η μετάβαση. Ολοκληρώνοντας, θα σταθώ στην ε, ευρωπαϊκή διάσταση. Είδαμε ήδη τις ε, ροές που παρατηρούνται και την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η Ευρώπη λοιπόν θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς για τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και για, τα, ε, για την παγκόσμια κοινότητα αλλά γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η θεσμική συνοχή αλλά και να υπάρχει συνεκτική πολιτική, η οποία θα ε, είναι επίσης συνεκτική και με τις ε, πολιτικές των επιμέρους χωρών. Όπως ε, πρότεινε και ο Επίτροπος Τίμερμαν στην έκθεση μας παρουσίασε. Μετά, ε, σε ό,τι αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ε, προωθήσουμε και σε άλλα σημεία του κόσμου. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει αντίκτυπο παγκόσμιο και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα, που βοηθούν ως προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικά για ε, τους στόχους που αφορούν το κλίμα αλλά και για την ε, αλλαγή χρήση της γης ε, που έχει επηρεάσει τη βιοπικιλότητα και τα οικοσυστήματα εν γέννη, δηλαδή παραγωγή τροφίμων κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει ε, ενδελεχής ανάλυση αυτού του σκέλους. Τέλος, να πω πως συνεργαζόμαστε με τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από τη συνεργασία αυτή έχει φανεί πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία για να εντοπιστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε λοιπόν τόσο με επενδυτές όσο και με τις επιχειρήσεις, με τους υπεύθυνους πολιτικής. Κάναμε ήδη ένα εργαστήριο, το πρώτο, όπου είδαμε ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως, πως χρειάζονται εργαλεία, χρειάζεται πλαίσιο για να καλυφθούν οι ελλείψεις. Στο μέλλον, λοιπόν, χρειάζεται να βοηθήσουμε την ε, επιστημονική έρευνα έτσι ώστε να, γι... να μην χάσουμε αυτήν την πολύ σημαντική ευκαιρία. Να συνδεθεί επίσης ή, ε, να συνδεθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης με την χρηματοδότηση και να δημιουργηθεί μια παγκόσμια διακυβέρνηση και διαχείριση αυτών των ροών έτσι ώστε να διαχειριστούμε καλά αυτήν την ε, μετάβαση. Χρειάζεται λοιπόν να εντοπιστούν οι συνθέσεις, ε, να αναπτυχθεί η επιστημονική έρευνα σε όλο τον κόσμο. αυτά λοιπόν ε, από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή και με τα χαρά να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, αν θέλετε λάβετε το λόγο για ερωτήσεις για τις δύο μελέτες. Μια ήταν μελέτη, η άλλη ήταν έκθεση που παρουσιάστηκαν. Και μετά όλοι οι ομιλητέ θα κληθούν να δώσουν απαντήσει, να αντιδράσουν στα σχόλιά σα. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, κύριε Κάλαμπαχ, έχει το λόγο. Σύντομη ερώτηση προ την πρώτη μελέτη. Θα δοθεί συνέχεια όσον αφορά την αναχώρα εξέλιξη για τα θέματα αυτά. Θα ήταν ενδιαφέρον κάτι τέτοιο σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Τίμερμανς στην αρχή. Να δούμε ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάισνερ. Και εγώ, σύντομότατη ερώτηση. Μπορούμε να βρούμε τις εκθέσεις κάπου, αυτές που, αυτή που παρουσιάστηκε στην τελευταία ομιλία. Έχουμε ένα αντίγραφο. Because... Όχι ακόμα. Ήταν δύσκολο να δούμε στον πίνακα στις οθόνες. Βλέπετε γι' αυτό. Ah, σας δώσουμε τις διαφάνειες. Την έκθεση την ίδια βλέπουμε, κύριε Λάινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις δύο παρουσιάσεις. Η Φιλανδία αναφέρεται και στο θέμα αυτό της δέσου επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Και είπατε ότι θέλετε να πρέπει να αναδιοργανωθούν οι προσεγγίσεις για τη δέους επιμέλεια. Είναι έτοιμε οι επιχειρήσεις. Οι κοινωνικοί παράγοντες θα ενταχθούν. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ληφθεί υπόψη και το θέμα του περιβάλλοντος και να τεθούν νομικά δεσμευτικά πλαίσια. Κάτι που προτείνει ο ΣΑ. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Κυρία Μακάβαν, ερώτηση. Μια εξήγηση θέλω. Αυτή η μελέτη τη καθηγήτρια Φούλμαν έχει ετοιμαστεί, παρουσίασε η καθηγήτρια Φούλμαν, ετοιμάστηκε για το Σεπτέμβριο, του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων, που το Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη θα εξετάσουν την προηγούμενη τετραετία. Γι' αυτό ετοιμάσατε τη μελέτη, έτσι. Είναι πάρα πολύ τεχνική. Ποια είναι τα βασικά μηνύματα που θα απευθυνθούν προς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και απορρέουν από τη μελέτη. Και η πρώτη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, είχε πολλέ λεπτομέρειες. Ε, που το τμήμα η διεύθυνση πολιτικής ανέθεσε. Θέλουμε να ξέρουμε ποιες, τι κάνουν τα κράτη-μέλη, ποια πάει καλά, ποια δεν πάει καλά. Ξέρω ότι είναι παριστάμενες και ΜΚΟ. Για το κλίμα δίνουμε επίσης ε, βραβεία, βραβεία για την καλύτερη επίδοση, για τη χειρότερη επίδοση. Ίσως και για τους στόχους αυτούς της βιώσιμης ανάπτυξης να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, για να υπάρχει παρακολούθηση και υποπτία. Μόνο η πολιτική πίεση θα σπρώξει κυβερνήσει να ακούσουν και να πιεστούν για να πετύχουν αποτελέσματα όσον αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Κυρία Χόιμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καθηγήτρια Φούρμαν, αναφέρατε <clears throat> ότι δεν είναι μόνο θέμα περιβάλλοντος και κλίματος, αλλά τίθενται και κοινωνικά θέματα. Αναφερθήκατε στις ανισότητες και τις ε, κοινωνικές αδικίες. Και είπατε ότι υπάρχουν και πισοδρομήσεις, ε, ανάπτυξη του εθνικισμού και του λαϊκισμού. Τα αντιμετωπίζετε ισότιμα στην έκθεσή σας. Τα θέματα περιβάλλοντος, για παράδειγμα, και κλίματος. Σε σχέση με τα άλλα, εάν ε, θέλουμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας Πρέπει παράλληλα να επιλύσουμε και τα κοινωνικά προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές αδικίες, ανισότητες ε, μεταξύ κοινωνιών, εντός των κοινωνιών. Πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε και με αυτό. Και πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό που είπατε, ότι δεν έχουμε μόνο ε, προκλήσεις σε επίπεδο πλανητικό, αλλά και προκλήσεις σε επίπεδο κοινωνικό να αντιμετωπίσουμε. Πολύ σπάνια έχω ακούσει τέτοιες διαπιστώσεις και νομίζω ότι είναι απίστευτα σημαντικό. Μήπως μπορείτε να πείτε τίποτα περισσότερο γι' αυτό παρακαλώ. Καλώ. ευχαριστώ πολύ. Καλό τους φιλοξενούμενους μας να απαντήσουν στις ερωτήσεις, να σχολιάσουν αυτά που υπόθηκαν. Κοιτάξτε, καταρχάς υπήρξε μια ερώτηση για τη συνέχεια που δοθεί. Αυτή ήταν η αρχική μου έκκληση. Όταν ξεκίνησα, αυτό είπα. Είναι αφετηρία αυτή. Είναι η βάση. Ένα εγχειρίδιο είναι αυτό. Έτσι σχεδιάστηκε. Όλοι από κάθε χώρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το έγγραφο και να έχουν μια βάση. Προχωρήσαμε πιο πέρα. Δεν περιγράψαμε μόνο την κατάσταση. Είναι περιγραφικοί οι πίνακες, αλλά έχουμε φεύγει αυτό που η αυτό τον τρόπο αξιολόγησης και τα διαγράμματα με τις χώρες και έχουμε και μετά αυτά τα μίνι διαγράμματα τα κυκλικά που είναι σαν και με τα... για τις επιδόσεις των χωρών. Βλέπουμε τι έχει σχεδιαστεί, ποιοι στόχοι έχουν θετεί. Έχουμε απεικονίσει την τρέχουσα κατάσταση, τι έχει σχεδιαστεί, τι έχει επιτευχθεί, ποιες μέθοδοι έχουν ε, ακολουθηθεί. Δεν έχουμε αξιολογήσει ακριβώς τι έχει ε, λειτουργήσει. Αυτή είναι η δεύτερη πτυχή που πρέπει να αναλυθεί. Θέλαμε όχι μόνο να δούμε στοιχεία, αλλά να έρθουμε σε επαφή με διαφόρους εκπροσώπους, να δούμε τι λεπτομέρειες υπάρχουν, τι απόψεις έχουν, τι εφαρμόσει στην πρακτική, τι μπορεί να υλοποιηθεί σε σχέση με το σχεδιασμό και μια πρόχειρη αξιολόγηση γίνεται. Χρειάζεται διεύρυνση, το είπε και η Λίντα να καλυφθούν περισσότεροι εμπλεκόμενοι. Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων εξέφρασαν άποψη. Πρέπει να γίνει αντιπαράθεση με τις απόψεις άλλων εμπλεκομένων και να δούμε πόσο εύρυθμα ε, προχωρούν όλα και να μάθουν οι μένα από τους δε. Σε κάποιο βαθμό αυτό ισχύει, αυτά συμβαίνουν. Αλλά εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να προσπαθήσει να συστηματοποιήσει τις προσπάθειες να προωθήσει τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης και εκμάθησης από ομοτήμους. Έχουμε μια μελέτη. Αυτή είναι η βάση για τη διακυβέρνηση, για τη θεσμική αντίδραση έναντι του θεματολογίου του 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ακούσαμε ερωτήσει προ τον Φραν Τίμερμαν, πώ θα κινηθεί η Μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητείται σε επίπεδο κοινοβουλίου, σε επίπεδο ΜΚΟ, σε τομεακό επίπεδο Χρειάζεται λοιπόν να εξεταστούν οι διάφοροι φορείς και διάφοροι τομείς. Να έχουμε όμως μια γενική εικόνα των προσπαθειών θέλουμε. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων για να προωθηθούν οι στόχοι. Χρειάζεται προώθηση, συστηματοποίηση της προσπάθειας. Μια στρατηγική θα ήταν καλή ιδέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά να δούμε βάση αρμοδιοτήτων ποιος αναλαμβάνει τι, ποιους στόχους πετυχαίνει, ποιους όχι. Χρειάζεται όμως στρατηγική. Είναι ένα εργαλείο στρατηγική. Εργαλείο για διαχείριση της προσέγγισης της διατομιακής με κάλυψη όλων των επιπέδων και όλων των φορέων. Πρέπει να δοθεί συνέχεια. Να υπάρξει κοινή προσπάθεια είχα αναφερθεί στην προσέγγιση των 28 χωρών τη ευρωπαϊκή Ενώσεω. και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ετοίμασε ανάλυση αναχώρα και πώς συμμετέχουν διάφορα εμπλεκόμενοι στι 28 χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα μπορούσε να υπάρξει και μεταξύ θεσμικών οργάνων συνεργασία και να συνεχιστεί η προσπάθεια της ΕΟΚΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια απάντηση. Ευχαριστώ. Ναι. Πρώτον, ε, χρειάζεται να ασκηθεί πολιτική πίεση. Συμφωνώ. Για παράδειγμα, έχουμε τη συνάντηση κορυφή για του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη το Σεπτέμβριο. Θα είναι κρίσιμη στιγμή για το πώ πάνε οι στόχοι αυτοί. Όπω ξέρετε, δεν αναλαμβάνει κανεί ε, την ηγεσία σε πλανητικό επίπεδο. Οπότε τότε θα κριθεί εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο πρωτοπόρου γιατί εάν οι στόχοι αυτοί θα αναφερθούν από τα μέσα και τα Και, και ε, να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό χάσμα. Ναι, σε κάποιες χώρες κάτι έχει γίνει, αλλά σε πολλές χώρες ακόμη δεν έχουν γίνει αρκετά και ιδίως από θεσμικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο, ε, από την θεσμική και κοινοβουλευτική πλευρά. Και τώρα ο κύριος ε, Βαν Πέτερσελ. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Πότε θα σας στείλουμε την έκθεση. Έχετε ήδη τις διαφάνειες. Η έκθεση θα ολοκληρωθεί ένα πρώτο σχέδιο τον Απρίλιο και το τελικό σχέδιο θα υποβληθεί το Σεπτέμβριο σε αυτή τη συνάντηση υψηλού επίπεδου στην ε, Νέα Υόρκη. Δεύτερον, ποια είναι τα κύρια μηνύματα που προκύπτουν από την έκθεσή μας. Θα επιχειρήσω να τα περιγράψω και σίγουρα η Εύα θα συμπληρώσει. Πρώτον, η έκθεση αυτή δεν στοχεύει να υποκαταστήσει τις ετήσιες εκθέσεις που δυστυχώς έχει το ίδιο όνομα GSDR, Παγκόσμια Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τα Ηνωμένα Έθνη δημοσιεύουν μια τέτοια έκθεση κάθε χρόνο που εξετάζει την εφαρμογή κάποιων από αυτούς τους στόχους. Η έκθεσή μας λοιπόν δεν υποκαθιστά αυτές τις εκθέσεις. Η έκθεσή μας είναι η πρώτη τετραετής έκθεση. Και στόχος μας είναι να πάρουμε λίγο περισσότερη απόσταση για να δούμε τι συστάσεις μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, να διευκολύνουμε την ε, επίτευξη συνολικά και των 17 στόχων κατά τις επόμενες ε, περιόδους. Τώρα, ένα βασικό μήνυμα. Πολλοί από αυτούς τους στόχους ε, δεν τα πάνε καλά. Δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς η έκθεσή μας, δεν κοίταξε αναλυτικά πώς εφαρμόζεται ο κάθε στόχος. Όπως είπα, δεν υποκαθιστά τις άλλες αυτές αιτήσεις εκθέσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, βασικό μήνυμα. Η ανθρωπότης δεν θα επιτύχει αυτούς τους στόχους μέσω ε, μικροαλλαγών, μικροπροσαρμογών ε, εδώ και εκεί. Όχι, χρειάζεται μετασχηματισμός. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη μετασχηματισμός στην έκθεσή μας. Και εξηγούμε τι σημαίνει μετασχηματισμός. Και για να επιτευχθεί αυτός ο μετασχηματισμός. Όπως είπε και η Εύα, τονίζω και εγώ, Πρέπει να ε, έχουμε άλλη προσέγγιση σε σχέση με τα συστήματά μας για να επιτευθούν οι πολλές απαραίτητες συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων μεθόδων για να έχουμε απτά αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των στόχων. Και υπάρχουν και πολλές δυνατότητες που προκύπτουν, που θα προκύψουν μέσω αυτών των συνεργασιών. Βεβαίως ε, ε, πρέπει να γίνουν κάπου αντισταθμίσεις, αλλά θα προκύψουν πολλές ευκαιρίες. Τις ευκαιρίες αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Έτσι απαντάω πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν, που ρωτήσατε. Άλλο μήνυμα βασικό που θέλω να δώσω. Την περιβαλλοντική πλευρά των βιώσιμων στόχων δεν θα την επιτύχουμε αν δεν εργαστούμε περισσότερο για το κοινωνικό θέμα. Είδατε τι έγινε με τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία πριν από μερικέ εβδομάδε. Ε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Λαμβάνονται περιβαλλοντικά μέτρα χωρίς όμως να εξεταστεί η κοινωνική επίπτωση. Τότε η κοινωνία δεν τα στηρίζει και δεν προωθούνται. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις ανισότητες και εντός και μεταξύ χωρών αν θέλουμε να υπάρχει ελπίδα επίτευξη αυτών των στόχων. Και τελευταίο βασικό μήνυμα ή ένα από τα τελευταία βασικά μηνύματα. Η συμβολή τη επιστήμης. Φυσικά οι 15 συντάκτε είναι επιστήμονες. Άρα ευλογάμε τα γένια μας, αλλά ίσως μέχρι στιγμή δεν έχει αξιοποιηθεί η επιστήμη όσο θα έπρεπε. Αν θέλουμε να αξιοποιηθεί πλήρως η τεράστια επιστημονική γνώμη, ε, γνώση συγγνώμη, που έχει επιτευχθεί από πολλούς επιστήμονες σε πολλά μέρη του κόσμου και να γίνουν αναγκαίες συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων αποτελεσμάτων αυτής της επιστημονικής έρευνας. Υπάρχουν τρόποι για να το επιτύχουμε. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά μηνύματα. δεν ξέρω πώς η Εύα θέλει να συμπληρώσει. Όχι, δεν έχω πολλά να πω. Πολύ καλά τα είπατε. Αλλά όλα αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος είναι πολύ ε, στενά συνδεδεμένα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης, για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γίνει μετασχηματισμός των συστημάτων. Το σύστημα, για παράδειγμα, παραγωγής και διανομής τροφίμων. Πρέπει να το δεις ε, και από πλευράς περιβαλλοντικής, από πλευράς κοινωνικής, όλες τις πλευρές. Η έκθεσή μας ακριβώς έτσι έχει δομηθεί. Αναφέρθηκα στη σχέση, της διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορών πλευρών του θέματος. Αλλά μπορεί όσοι επιχειρούν να ε, βελτιώσουν λοιπόν την κατάσταση να ε, επινοήσουν νέες συνδέσεις. Και το θέμα της δέουσας επιμέλειας από πλευράς επιχειρήσεων. Μπορούν οι επιχειρήσεις να διεξαγάγουν τη δέουσα επιμέλεια. Πολλέ επιχειρήσει το γνωρίζω, δεν ασχολούνται καν με αυτό. Αλλά υπάρχουν και αρκετέ που είναι πρωτοπόρε ε, στα θέματα αυτά. Και υπάρχουν συστήματα τα οποία υπερβαίνουν τα εθνικά όρια. Βλέπω λοιπόν φως στο βάθος της σύραγγας. Πρέπει λοιπόν πολλά να κάνουμε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, όλοι ξέρετε πρέπει να συμμετέχουν. Όλοι οι επιστήμονες, παγκόσμια. Και να αλληλοβοηθούνται. Δεν είναι μόνο θέμα χρηματοδότησης της έρευνας, αλλά και δικτύωσης υποδομών αλλά κυρίως πρέπει να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Ένας συνάδελφος ε, είναι από την Ιαμαϊκή, ε, αλλά είναι καθηγητής και στο Λονδίνο. Μόνο όταν είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τώρα για την έκθεση. Ενημερώναμε σε κάθε φάση εκπόνησής της ε, τι έχουμε επιτύχει και προς τα που πηγαίνουμε. Όλα λοιπόν ε, όσα σας δείξαμε είναι πάντα εν εξελίξη. Θα δημοσιευθεί αργότερα, αλλά θέλαμε ήδη να τα μοιραστούμε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για την παρουσίαση. Ο λόγος πίσω στην κυρία Μακάβαν. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τι μελέτε, Είναι πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία και θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη θητεία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόζει το έγγραφο προβληματισμού. Αλλά και θα βοηθήσει όσου επιστρέψουν και συμμετασχούν σε ακροάσει και στο έργο της Επιτροπής. Ε, η κυρία Βαλεάν πρέπει να φύγει, οπότε θα την αντικαταστήσει ο αγαπητός αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ. Ζήλ, χαιρόμαστε που σε βλέπουμε και περνάμε ευθύ αμέσως στο δεύτερο μέρος της ακρόασης με την ε, ομιλία του Τζέφρι Σάξ, πρόεδρου του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και διευθυντή του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ε, Τζέφρι, προσπάθησε εδώ και χρόνια να συνδέσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ε, την έρευνα. Σήμερα ακούσαμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βάλει ακόμα πιο ψηλά ε, στις προτεραιότητες της, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ενημερώθηκαν και οι συνάδελφοι που δεν γνώρισαν για τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών ότι κάθε χρόνο το δίκτυό σας δημοσιεύει έναν πίνακα επιδόσεων για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να δούμε ε, που βαδίζουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε από τη Νέα Υόρκη μέσω της Ουάσιγκτον. Σήμερα το πρωί λοιπόν φτάσατε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας δίνω μέσα στο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι εκπληκτικό ε, το ότι υπάρχουν όλες αυτές οι εξελίξεις, έχει σημειωθεί τόση πρόοδος ε, εδώ στα θεσμικά όργανα. Είναι πολύπλοκη η διαδικασία και είναι λοιπόν ε, εκπληκτικό το ότι δουλεύουν όλα έτσι όπως ε, θα έπρεπε και όπως είπατε σήμερα το πρωί όλα συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει διατομεακή διάσταση, μακροπρόθεσμη πολιτικά, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι πρόκειται για προγράμματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα 30-40 ετών. Και αυτός ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας ε, έχει θεσπιστεί σε μια περίοδο πολύ φορτισμένη πολιτικά. Συντελούνται αλλαγέ ε, λοιπόν που είναι αναγκαίε και η διαδικασία αυτή απεδείχθη πω ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έχει έρθει όμω ε, η στιγμή που συμπληρώνεται ένα τέταρτο του αιώνα, 25 χρόνια από την ε, Σύνοδο Κορυφή για το Κλίμα και η πορεία που ακολουθείται δεν έχει αλλάξει πολύ. Βλέπουμε ότι η κακή, ας πούμε, εντό αγωγικών συμπεριφορά δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ, όμως ε, η κλίμακα και η τάξη μεγέθους ε, αλλάζει. Έχουμε λοιπόν επιβάρυνση του πλανήτη είτε περιβαλλοντικά είτε κοινωνικά η οποία είναι ε, επιβάρυνση που προκαλεί ο άνθρωπος. Με τρομερές ε, επιπτώσεις, αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα με αύξηση των ε, ανισοτήτων σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Και αυτό νομίζω δείχνει εν μέρη πόσο ισχυρά είναι τα συμφέροντα πίσω από αυτές τις αλλαγές και πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία να δημιουργηθεί ε, μια παγκόσμια, ένα παγκόσμιο πλέγμα που θα, που θα συνδέει όλον τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν πως οι καιροί αλλάζουν ταχύτατα, από την άλλη προχωράμε πολύ γρήγορα και είμαστε κοντά στο χείλος του γκρεμού. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή λοιπόν για να μην πέσουμε. Αν δείτε στο χάρτη στον παγκόσμιο χάρτη ποιε χώρες είναι πολύ κοντά στο να πετύχουν τους στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, ε, θα δείτε πως στην κορυφή βρίσκονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα και της Ευρώπης γενικότερα. Αυτό είναι καλό, διότι θα έλεγα πως οι αξίες, τα κίνητρα και η πολιτική στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο κοντά σε αυτούς τους στόχους σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Στις Ηνωμένε Πολιτείες, για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί επιτάχυνση, αλλά προς την άλλη κατεύθυνση. Μεγιστοποιείται η ανάπτυξη τεχνολογίας για τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Υπάρχουν οι σχετικοί ε, κανονισμοί οι οποίοι ε, σε συνδυασμό με τον ε, πρόεδρο, ο οποίος είναι τελείως αντίθετος στους στόχους του για την προστασία από την κλιματική αλλαγή δεν βοηθάει. Δεν θα τον πω ψυχοπαθή, αλλά θα περιοριστώ στο ότι είναι αντίθετο. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι αναλύσει γίνονται ακόμα σε εθνικό επίπεδο κατά κύριο λόγο. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο, το τι γίνεται, γιατί το κάνουμε, τι δεν κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως οι προσπάθειες αυτές δεν ε, γίνονται συστηματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δηλαδή να υπάρχουν μεμονωμένες ε, έρευνες, μεμονωμένες μελέτες και να μην υπάρχει από κοινού μία έρευνα, ε, μία προσπάθεια από την Ευρώπη των 27, α πούμε των 28. Όλες οι προτινόμενες λύσεις θα πρέπει να είναι λύσεις μεγάλης κλίμακας γεωγραφικής και πληθυσμιακής. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτόμαστε μεγαλόπνοα ε, και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στις επιμέρους χώρες, διότι τα συστήματα μεταφορών, τα ενεργειακά ε, συστήματα είναι συστήματα ε, που συνδέονται μεταξύ τους και δεν είναι ένα πάζλ με την κάθε χώρα να αποτελεί ένα κομμάτι. Χρειάζεται ένας συνδυασμός προσπαθειών έτσι ώστε να σημειωθεί πρόοδος. Βέβαια, Χρειάζονται και οι τοπικές λύσεις, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε την ε, διασυνδεσιμότητα και την ε, παγκόσμια διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να χαράξει μονοπάτια τα οποία θα βοηθήσουν κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ε, διαφαίνεται πολύ. Όμως είναι πιο μπροστά από όλα τα υπόλοιπα κράτη, από όλε τις άλλες περιοχές του κόσμου, τόσο σε μια πολιτική πολύ συνεκτική, ε, αλλά και ως ε, προς ε, τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν. Νωρίτερα φέτος δημοσιεύσαμε μία έρευνα για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Θα τους αναφέρω λοιπόν συνοπτικά. Υγεία, εκπαίδευση, ενέργεια, επισητισμός, πόλης και ε, τεχνολογία της πληροφορίας. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδί. Για το 2019 ε, και, η, και εσείς έχετε παρόμοιες ε, προτάσεις, όμως είναι πολύ σημαντικό να δούμε πως αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν με πάρα πολύ δουλειά. Χρειάζεται προσπάθεια για την τυποποίηση, για την ε, οργάνωση, για την εφαρμογή. Ε, δεν θα σταθώ τόσο πολύ στην υγεία και στην εκπαίδευση, αλλά για την ενέργεια. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μέχρι τα μέσα αυτού του αιώνα πρέπει να αποδεσμευτούμε τελείως από τη χρήση άνθρακα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει αυτό μέσω ενός ε, δικτύου που θα τυποποιήσει ε, το ενεργειακό δίκτυο. Δηλαδή να συνδεθούν όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, να συνδεθεί η Ευρώπη με την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, να ε, πετύχουμε το στόχο της μηδενικής παραγωγής άνθρακα και να μην αφήσουμε αυτό να το λύσει κάθε χώρα μόνη της. Να είναι μια συντονισμένη ομαδική προσπάθεια. Ο συντονισμός είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός και η αποκέντρωση. Ακριβώς διότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ε, πηγές που παράγονται εξεχωριστά είναι πολύ σημαντικό να τις ε, συνδέσουμε, διότι ο ήλιος δεν ε, σε όλη την ε, επικράτεια της Ευρώπης, δεν έχουμε λιακάδα κάθε μέρα, υπάρχουν συννεφιές, υπάρχουν βροχές, γι' αυτό και χρειάζεται ένα πλέγμα, ένα δίκτυο στο οποίο θα συνδέονται όλες οι ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Κάτι το οποίο μας λείπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Πού είναι ο χάρτης. Να δούμε, να δούμε το χάρτη, να δούμε και τη Γερμανία η οποία έχει ενεργειακή πολιτική, την οποία εφαρμόζει για 8η ε, χρονιά, μας ε, λέει ότι μέχρι το 2038 έχει σκοπό να ε, σταματήσει την χρήση άνθρακα ως καυσίμου. Αυτές οι αλλαγές είναι κομμάτι ενός σχεδίου με ορίζοντα 20-30 ετών, το οποίο σχέδιο θα πρέπει να προσαρμοστεί φυσικά ε, σε βάθος χρόνου, όμως ε, είναι ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο που λείπει. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι δεν μπορείς να αλλάξει σε μία νύχτα τα πάντα. Είναι μία αλλαγή που θα γίνει βήμα-βήμα, θα γίνει σε στάδια, έτσι ώστε να φτάσουμε στην αποδέσμευση των άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα. Χρειάζεται να συμμετέχουν όλοι. Και ε, η παραγωγή ενέργειας και η βιομηχανία και ε, οι επιχειρήσεις. Δεν μπορεί καμία χώρα να το καταφέρει αυτό μόνη της. Χρειάζεται συνεργασία. Έπειτα, από την πλευρά της παραγωγής τροφίμων τώρα, το ζητούμενο είναι να παράγονται τρόφιμα ε, περιβαλλοντικά βιώσιμα και ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μία λοιπόν έχουμε τα τρόφιμα που παράγονται στην Ευρώπη και τα εισαγόμενα τρόφιμα διότι καταστρέφεται ο Αμαζόνιος, καταστρέφεται το αρχιπέλαγος της ε, Ινδονησίας, είναι ο χάρτης που βλέπατε πιο πριν στην παρουσίαση για τις ε, διασυνδέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη έχει τεράστια ευθύνη και τεράστιο ρόλο ε, στην διασφάλιση αυτής της συνοχής. Δεν υπάρχει ακόμα ένα παγκόσμιο σχέδιο, όμως Τις τελευταίες εβδομάδες δημοσιεύτηκαν ε, δύο μελέτες ε, για το θέμα αυτό. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα η μία από αυτές, η οποία οδηγείται σε ένα βασικό συμπέρασμα, ότι χρειάζεται να αλλάξει η διατροφή και η παραγωγή τροφίμων προς μια πιο βιώσιμη μέθοδο παραγωγής και κατανάλωσης τόσο κρέατος όσο και μη ζωικής πρωτεΐνης. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο ε, που τρεφόμαστε και να, ε, να αξιολογούμε διαφορετικά την ε, αλυσίδα αξίας. Χρειάζεται λοιπόν κατεύθυνση και νομίζω πως η μελέτη το δείχνει αυτό. Θεωρώ λοιπόν πως είναι σημαντικό πρώτον να αναβαθμίσει η επόμενη Κομισιόν ε, το σχέδιο αυτό, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι μεγάλες ε, αλλαγές και μεταβολές. Φυσικά να επιτευχθεί η συνοχή σε όλα τα κράτη-μέλη ε, και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών. Και να τονίσω ξανά ότι χρειάζεται δράση σε υψηλό επίπεδο. Δεν μπορούμε να χαράξουμε ε, αυτή την πολιτική και τα μονοπάτια από, πάνω, από κάτω προς τα πάνω. Χρειάζεται το αντίθετο. Χρειάζεται να έρθει από ψηλά. Και αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θα έδινα έμφαση στην ε, ενεργειακή μετάβαση. Σαν έναν απλό στόχο δηλαδή. Αποδέσμευση από άνθρακα. Από τον άνθρακα. Σύντομα. Έπειτα αλλαγή στη χρήση της γης προς περισσότερη βιοπικιλότητα προς ε, περισσότερα βιώσιμα τρόφιμα. Επίσης, δεν έχουμε περιθώριο στην Ευρώπη για να καλλιεργήσουμε βιοκαύσιμα. Αν δείτε την ε, ισορροπία των οικοσυστημάτων θα παρατηρήσετε ότι η ε, πολιτική που ακολούθησαν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα βιοκαύσιμα ήταν λάθος. Δεν έχουμε αρκετή γη, δεν έχουμε αρκετό νερό έτσι ώστε να ε, χρησιμοποιήσουμε τα οικοσυστήματα για να καλλιεργήσουμε τόσο τρόφιμα όσο και βιοκαύσιμα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, όλους τους διαθέσιμους πόρους, ακόμα και τις ερήμους. Τρίτον, επίσης σημαντικό είναι η περιφερειακή πολιτική στην Ευρώπη η οποία θα δημιουργήσει πρότυπα για αυτήν την ε, μετάβαση. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι περιφέρειες ε, με υψηλή ανεργία, με χαμηλό εισόδημα θα μπορέσουν να συγκλίνουν προς τις ε, υπόλοιπες. Πώς θα αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Είναι μια πολιτική η οποία φυσικά θέλει σχεδιασμό δεκαετιών και ήδη ακολουθείται, όμως χρειάζεται ενίσχυση. Επίσης υπάρχει και κάτι συμπληρωματικό θα έλεγα, ε, ο ρόλος δηλαδή της Ευρώπης. με τις αξίες της και με τον γενικότερο προσανατολισμό της η Ευρώπη ε, ηγήθηκε και θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μην χάσετε αυτήν ε, την ε, πρωτοκαθεδρία, αυτήν την ε, ηγετική ικανότητα και ηγετική θέση. Μην νομίζετε πως έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμα. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ουσιαστικό ρόλο αν θέλουμε να πετύχει το σχέδιο. Πρώτον, η αναπτυξιακή βοήθεια παραμένει ζωτική σημασίας. Και η αναπτυξιακή βοήθεια στην Ευρώπη πρέπει να, γίνει, πρέπει να συγκλίνει περισσότερο έτσι ώστε να συμφωνεί με αυτές τις ε, μεταβολές. Δεν πρέπει να είναι απλώς ένα άθισμα των 28 προγραμμάτων ε, βοηθείας. Θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Αυτή είναι η άποψή μου και καλύτερη και ισχυρότερη από ό,τι τώρα. Δεύτερον, ο ρόλος της Ευρώπης όσον αφορά τι αλλαγέ για το κλίμα. Θα πρέπει μέχρι το 2050 παρά για τον άνθρακα η Ευρώπη όπω η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλε περιοχέ του κόσμου. χωρί την ηγεσία τη Ευρώπη σε αυτό το τομέα δεν θα συμβεί αυτό. Χρειαζόμαστε ισχυρή συνεργασία με την Κίνα, με την Ινδία και αν ε, μπούμε σε ανόητους εμπορικούς πολέμους ή σε νέα πεδία μαχών, δεν θα πετύχουμε αυτή την συνεργασία. Υπάρχουν πολλά προσυζήτηση από αυτού. Η Κίνα έχει υπέροχες ιδέες για τις παγκόσμιες διασυνδέσεις σε ενεργειακό επίπεδο και θα πρέπει να έχουμε μια πράσινο, πράσινο δρόμο του Πεκίνου και η συμμετοχή της Ευρώπης. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν άλλες ιδέες Εμεί πολεμάμε με την Κίνα. Αυτή είναι μια άλλη ανόητη αμερικανική ιδέα τώρα. Παροτρύνω την Ευρώπη να μην ακολουθήσει παρόμοια κατεύθυνση, διότι θα τεθεί τέρμα έτσι στη δυνατότητα παγκόσμιας συνεργασίας που είναι ζωτική σημασία. στο τομέας, στον οποίο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, η Ευρώπη είναι στη διακυβέρνηση της τεχνολογίας πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε το σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια μας, τη διασυνδεσιμότητα τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι και πρόβλημα όμως ισότητας και ελευθερίας. Το GDPR και άλλα ε, θέματα ευαισθησίας στην Ευρώπη είναι σωστές προσεγγίσεις. Η Ευρώπη λέει πώς μπορούμε να έχουμε την ψηφιακή τεχνολογία χωρίς να έχουμε απώλεια ελευθεριών, χωρίς απώλεια ιδιωτικότητας και νομίζω ότι αυτό από πλευρά ε, θεματικής είναι κάτι σημαντικό για μια βιώσιμη αλλαγή και μεταμόρφωση. Πρέπει να έχει υψηλή ποιότητα. τέταρτο τομέα. είναι η διακυβέρνηση της όλη αλυσίδα αξιών. Αυτό δεν μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα με ανεύθυνες αλυσίδε αξιών. Είναι παγκόσμια προβλήματα και δεν έχουμε επιλύσει το πρόβλημα της διακυβερνήσεως αυτής της αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει ανευθυνότητα σε αυτήν την αλυσίδα, διότι οι επιχειρήσεις έχουν σχεδιαστεί για ανευθυνότητα. Περιορισμένη ευθύνη αποκαλείται αυτό. Στις ΗΠΑ Πολιτείες αυτό σημαίνει μπορούμε να παραβούμε τον νόμο όποτε θέλουμε, αλλά δεν σημαίνει απόλυτα αυτό σημαίνει ότι, ότι αν είναι εκτός της δικής μας εταιρικής συμπεριφοράς εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Αυτό για διασυνδεδεμένο κόσμο είναι κάτι που δεν μπορεί να βιώσιθει. Χρειάζεται διακυβέρνηση της όλης αλυσίδας των αξιών. Υγείται η Ευρώπη σε αυτό, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί η προσέγγιση εθελοντικά. Πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμοστεί, να υπάρχει επιμερισμός των ευθυνών για, όλη την, για όλο τον τομέα, για τη γεωργία, για τα ορυχεία, για την ενέργεια και ούτω καθεξής. Εν τέλει, θα ήθελα να πω, εν γέννη, ότι η συμπεριφορά των εταιριών και η φορολογική συμπεριφορά είναι σημαντικά στοιχεία. Ο ευρωπαϊκός προβληματισμός περί διακυβέρνησης των εμπλεκομένων και διαφερομένων τομέων είναι κάτι πολύ σημαντικό και ηγείται εκεί η Ευρώπη η ΕΠΑ τελικά προσπαθεί να βελτιστοποιήσει το κέρδος των μετόχων. Η ιδέα συνδιαχείρισης του τομέα των επιχειρήσεων στη ΣΥΠΑ είναι κάτι αντίθετο από την οτροπία που επικρατεί στη ΣΥΠΑ. Και είναι πολύ σημαντικό για τη βιώσιμη ανάπτυξη να ακολουθηθεί η ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η διαχείριση των επιχειρήσεων, ο τρόπος που κινούνται οι επιχειρήσει, να είναι ένα σημαντικό θέμα για το μέλλον είναι πολύ ουσιαστικό για, τις, για τους φορολογικούς ε, παραδείσους. Ε, υπάρχουν οι χειρότεροι φορολογικοί παράδεισοι στον κόσμο, στην Ευρώπη και ε, υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ των φορολογικών παραδείσων και εκείνοι που είναι κατά. Και αυτή η αντιπαράθεση σκοτώνει τη διαδικασία. Η φορολογική παράδειση είναι πολύ επιβλαβής για τα δημοσιονομικά. Όσο υπάρχουν μεγάλη φορολογική παράδειση, που δημιουργούνται αυτοί οι παράδεισοι από τι ισχυρέ χώρες, δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχου μας. Τέλος, κάποια λόγια για την όλη διαδικασία, τη διαδικαστική. Και αυτή είναι η ουσία της αλλαγή και της μεταμόρφωσης. Για τη διαδικασία να πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερο προπολογισμό, το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, για να πετύχει του στόχου τη. Νομίζω ότι μεγάλη πρόκληση για το 2020 ένας ευρωπαϊκός υπολογισμός που αυξάνεται σε ένα υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν μπορείτε να έχετε μια Ευρώπη κατά την αποψή μου που είναι ενωμένη με βιώσιμο τρόπο, με έναν προπολογισμό που είναι ενωμένη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη με τα επίπεδα σημερινά του ευρωπαϊκού προπολογισμού, πολύ χαμηλό. Μετά οι διάφορε ε, μήτρε υπολογισμών, οι δικτυώσει και υπολογισμοί πρέπει να έχει σωστή προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του υπολογισμού προσέγγιση επιτριμήνουν να ενημερώνει μέσω στοιχείων της Eurostat, να δίνει σαφή στοιχεία, να είναι όρατα. Τώρα καθημερινά έχουμε στοιχεία και δείκτες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Πρέπει να έχουμε πίνακες και γι' αυτό και για τη φτώχεια κλπ. Όλα αυτά είναι εφικτά. Μετά, θα ήθελα να προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πλησιάσει τα διεθνή κοινοβούλια, άλλα κοινοβούλια του κόσμου, να γίνονται, να διοργανωθούν ακροάσεις με συμμετοχή άλλων κοινοβουλίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κάθε κοινοβούλιο χρειάζεται αυτού του είδους τη συζήτηση. Πολύ εύκολο τώρα να υπάρξει διασύνδεση και μέσω διαδικτύου, μέσω των οθονών με τηλεδιασκέψεις και νομίζω ότι θα μπορούσατε να ηγηθείτε τέτοιων διασυνδέσεων. Τέταρτον, πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια βιομηχανική πολιτική που ταιριάζει με την οριστατική. προσωπικά. Εγώ ήμουν υπέρ τη συγχώνευσης Siemens Alstom διότι δημιουργείται έτσι φορέας τύπου ε, Airbus στην κλίμακα αυτή μεγάλη επιχείρηση στον τομέα υψηλής τεχνολογίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη πολύ σημαντικό για την αλλαγή που χρειαζόμαστε και, εν πάση περιπτώσει, χρειαζόμαστε μια βιομηχανική πολιτική που αναλογεί με την κλίμακα της μεταρρύθμισης που απαιτείται και που έχει δρομολογηθεί και που ταιριάζει και με την φύση της παγκόσμιας οικονομίας όπως διαμορφώνεται. Χρειάζονται μεταμορφώσεις διάφορες πορείες, διάφορες στατηγικέ, διάφορους ε, σχεδιασμούς ε, με προπτική 20 ή 30 ετή όχι ιδέες απλές και ευχολόγια. Χρειαζόμαστε χαρτογράφηση του προγραμματισμού, της πορείας, που θα είναι, για η παραγωγή της ενέργειας, πώς μεταδίδεται, που είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που υπάρχει βιοπικιλότητα, ε, πώς παράγεται η ενέργεια από βιολογικές πηγές. Τώρα δεν έχετε τέτοια χαρτογράφηση η Ευρώπη, ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε οι περισσότερες άλλες περιοχές του κόσμου. Λοιπόν, ε, αυτές είναι κάποιες διαδικασίες που ήθελα να περιγράψω και να τονίσω. Να κλείσω όπως ξεκίνησα. Αυτό είναι το δικό σας θεματολόγιο. Πιστέψτε με, αν η Ευρώπη δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, καμία άλλη περιοχή του κόσμου δεν θα καταφέρει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η Ευρώπη είναι πιο κοντά στη λύση από όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου. Ίσως να μην το βλέπετε έτσι, να μην το αισθάνεται κανείς σε το μέσο της πολιτικής διαμάχης, αλλά είναι η αλήθεια. Και η συζήτηση που άκουσα το πρωί, τότε που συζητούσατε τις εκθέσεις, είναι μια συζήτηση που δεν άκουγα ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι είπα τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω, ακόμα και αν λύσουμε τα πολιτικά μας προβλήματα. Απλώς μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Ήμουν στη Ουάσιγκτον χτες. Τώρα είναι δυνατόν για δύο χρόνια δεν μπορούσα να, να πατήσω πόδι στη Ουάσιγκτον. Ήταν πάρα πολύ οδυνηρό. Ακόμα είναι οδυνηρό. Τώρα τουλάχιστον οι δημοκράτες έχουν κάποιο έλεγχο του Κογκρέσου και, και ε, μπορούν να ελέγχουν κάπως τον ε, πρόεδρο που είναι επικίνδυνος και δεν ενδιαφέρεται καθόλου γι' αυτό. Μπορείτε εσείς να ηγηθείτε του θεματολογίου. Δεν πρέπει να ξεφύγετε από αυτό, να συνεχίσετε όχι μόνο προς όφελος της Ευρώπης, αλλά προς όφελο όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τζέφρι. Πρώτα απ' όλα μα έδωσε λόγου για να ελπίζουμε και να είμαστε χαρούμενοι γιατί πολύ συχνά αυτέ οι συζητήσει λένε δεν προχωράμε. Πάμε προ τα πίσω. Η Ευρώπη ηγείται αυτή τη προσπάθεια. Κρίμα που ο Επίτροπο Τίμερμαν δεν ήταν εδώ να ακούσει το μήνυμά σα για το ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την πρωτοπορία. Ούτω ώστε και κατά την επόμενη πενταετία που θα έχουμε νέο Κοινοβούλιο και νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνουμε κάτι. Έχουμε αυτό το έγγραφο προβληματισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρει εναλλακτικέ λύσει. Μόνο μία από αυτέ τι εναλλακτικέ λέει ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμένη ε, προσπάθεια να προωθηθεί το θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλε δύο για μένα παράδεκτε. Σήμερα λοιπόν είχαμε την ε, προηγούμενη εβδομάδα αυτό το έγγραφο προβληματισμού. Το Κοινοβούλιο θα αντιδράσει και θα υιοθετήσει μια θέση γι' αυτό πριν από τι εκλογέ για να υπάρχει θέση του Κοινοβουλίου πριν την ε, συζήτηση υψηλού επίπεδου το Σεπτέμβριο. Έχουμε λοιπόν υλικό μπροστά μας για να διαμορφώσουμε τη θέση μας και τα αιτήματά μας έναντι της Επιτροπής και έναντι των κυβερνήσεών μας, ούτως ώστε η Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση. Λοιπόν, τώρα διάφοροι έχουν ζητήσει το λόγο. Τέσσερις συγκεκριμένα. Πόσοι ακόμη θα ήθελαν το λόγο. Έχω Χάουταλα, Χόιμπουχ, Κάντμπαχ, Λίτς, αυτή. Πόσο χρόνο έχουμε, Ντανατέλα? 20 λεπτά, ωραία. Δύο λεπτά ο καθένας. Χάταλα. Ευχαριστώ πολύ για τις στρατηγικές σας συμβουλές και την εμπιστοσύνη σας ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα πάει καλά. Σημερίζουμε αυτήν την αισιοδοξία. Πείτε μας παρακαλώ λίγο περισσότερα για το πώς ε, θα έχουμε αυτήν την ε, δεσμευτική διακυβέρνηση της αλυσίδας αξιών. Γιατί γίνονται έντονες συζητήσεις εντός και γύρω από την Ένωση και εντός των κρατών μελών για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Κάποια κράτη-μέλη όπως η Γαλλία ήδη έχει ε, νομοθεσία για οριζόντια δέωση επιμέλεια που θα μπορούσε να είναι πρότυπο ε, που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι πεπισμένη ότι η νέα Επιτροπή θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια κουρελού ε, νομοθεσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έχει απλώς νομοθεσία κατά της ε, δουλείας, ενώ η Γαλλία είναι στο άλλο άκρο με την οριζόντια αυτή δέως επιμέλεια. Πώς μπορείτε να μα συμβουλεύσετε ιδιαίτερα για τις ε, μη βιώσιμες ε, ε, αλυσίδες. Τι μπορεί να κάνει η Ένωση για να παίξει ηγετικό ρόλο, αν καταφέρει να λειτουργήσει σωστά, θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια κατάσταση. Ευχαριστώ. Χάιντι. Η Μαρία Χόιμπουχ. Ε, όπως μου υποβλήθησαν τετήματα, δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εντάξει, μ' ακούτε, τώρα. Ωραία λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν έλεγα για την παρουσίασή σας. Τελειώνοντα, είπατε ότι η Ευρώπη ε, είναι πιο κοντά στη λύση. Μα χαροποιεί αυτό. Αλλά νομίζω είναι επικίνδυνο να λέμε τέτοια πράγματα. Γιατί εμεί εδώ ω Κοινοβούλιο έχουμε κάνει πολλέ συζητήσει για το θέμα αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε κατόπιν, είμαστε πράσινοι, είμαστε πιο φιλόδοξοι και ακούμε το αντεπιχείρημα, μα ήδη κάνουμε τόσο πολλά. Και χαίρομαι που είπατε επίση ότι πρέπει να χάσει τον ηγετικό τη ρόλο η Ευρώπη. Γιατί ορισμένε φορέ ανησυχώ ακριβώ για αυτό το ρόλο. Γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι μα ήδη τα πάμε πολύ καλά. Και ναι μεν ε, ε, είμαστε πρωτοπόροι αλλά δεν είμαστε πάντα συνεπείς. Για παράδειγμα για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Πρέπει να είμαστε συνεπείς εδώ. Για παράδειγμα Στη ημερήσια διάταξη θα ψηφίσουμε μία γνωμοδότηση για την επόμενη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Κάθε φορά που έχουμε νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, θέτουμε το πλαίσιο για τα τρόφιμα, που είναι μέχρι κλειδί. Και αποφασίζουμε λοιπόν την πορεία προς την επόμενη επταετία, δηλαδή μέχρι το 2027, 2021-2027 συγκεκριμένα. Και δεν είναι απλό να είναι κανείς φιλόδοξος. Γιατί από τη μία έχουμε τις μεγάλες ε, αγριοβιομηχανικές επιχειρήσεις, ε, από την άλλη μεριά θέλουμε υγιή τρόφιμα, διατήρηση του ε, εισοδήματος των γεωργών, σταθερότητα των αγορών, Δύσκολο να συνδυαστούν όλα αυτά. Και είναι κρίμα που δεν είναι πλέον παρόντες οι συνάδελφοι οι οποίοι εδώ ε, θέλουν να φρενάρουν την πορεία μας. Και αναφέρω τα τρόφιμα γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα από, προ, από πλευράς προοπτικής ΔΕΒΕ αλλά και από πλευράς Άγκρη. Εγώ ίδια είμαι γεωργός. Και θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε και στι εκμεταλλεύσεις και στην πολιτική για να υπάρξει αυτός ο μετασχηματισμός. Πρέπει να σταματήσει η κατανάλωση κρέατο. το ξέρουμε αυτό. Αλλά εμείς οι πράσινοι πριν από, μερικές, ε, πριν από μερικά χρόνια αποτύχαμε ιδιαίτερα όταν έγιναν ε, εκλογές στη χώρα μας, όταν είπαμε ότι μία μέρα τη βδομάδα σε, ε, σε όλα τα δημόσια εστιατόρια και καντίνες να υπάρχουν μόνο φυτοφαγικά ε, εδέσματα. Ήταν μια προσπάθεια. Έχετε ιδέες ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, προωθήσουμε περισσότερο ακριβώς αυτή την ιδέα των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην κατανάλωση τροφίμων. Γιατί η ενέργεια και τα τρόφιμα είναι Τομείς κλειδί. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα σχέδιο πορεία. Εάν το κάνουμε αυτό σε αυτούς τους τομείς, νομίζω ότι θα τα πάμε καλύτερα και σε άλλους τομεί. Ευχαριστώ Μαρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνεται εκθετικά αυτή τη στιγμή ο αριθμός των ατόμων που είναι φυτοφάγοι ή και vegan. 28% είναι η γενιά των ε, παιδιών της χιλιετίας. Τους ανέφερε και ο Επίτροπος Τίμερμα σήμερα το πρωί. Είναι ενδιαφέρον ότι μπορεί να γίνονται πραγματικά τρομερές αλλαγές μετασχηματισμοί στις ε, συνήθειες. Όλο και περισσότεροι βλέπουμε είναι, όλο και περισσότεροι είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Η Κάρεν Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα Πολύ ενδιαφέρουσα και πλευρή η παρουσίασή σας. Είδαμε πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Ναι, μεν κινούμεθα προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αρκετά γρήγορα. Και χαίρομαι και για τα θετικά σας πορίσματα. Λοιπόν, καταρχάς να διαπιστώσω κάτι. Είπατε ότι δεν γίνεται τέτοιου τύπου συζήτηση στι Πολιτείε. Είπατε ότι αν υπήρχαν εκπρόσωποι όχι, εγώ να σας πω ότι εάν ε, είχαμε εδώ προσώπους από όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου θα ήταν πολύ διαφορετική συζήτηση. Εμείς εδώ είμαστε δεσμευμένοι ιδιαίτερα για να επιτύχουμε τους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης κτλ αλλά δεν είμαστε πλήρως αντιπροσωπευτικοί συνολικά για το Κοινοβούλιο. Αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά. Όταν υποβάλλουμε πολύ φιλόδοξες προτάσεις ω ΕΝΒΙ και στην Ολομέλεια, Πολλέ από αυτές τις προτάσεις δεν περνάνε. Επιτυγχάνουμε ορισμένα πράγματα και είμαι περήφανη για όσα έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια ως Κοινοβούλιο, αλλά διαπιστώσαμε ότι κάθε δράση προκαλεί αντίδραση. Υπάρχουν έντονες ε, και θορυβώδεις αντιδράσεις πολλές φορές. Όταν θέλουμε να υπάρξει ένα πλαίσιο για βιώσιμη οικονομία, τότε υπάρχουν αντιδράσεις που βασίζονται στο βραχυπρόθεσμο κέρδος. Είναι γενικά κοντό, κοντόθωρες, δεν ενδιαφέρονται για το μακρόπνο μέλλον. Και κάτι άλλο που υπόθηκε είναι πολύ ενδιαφέρον ότι θα πρέπει και τα 28 κράτη-μέλη να έχουν διακυβέρνηση για την εφαρμογή των ε, βιώσιμων στόχων. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι τα πάνε καλά τα κράτη-μέλη. Διότι κάποιες ε, αξιολογήσεις κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν είναι τόσο ενθουσιώδεις. Ερώτημα λοιπόν. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοντόθαρες θεωρήσεις που ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος. Πώς μπορούμε λοιπόν να τις αντιμετωπίσουμε μέσω της επιβολής των δικών μας μακροπρόθεσμων βιώσιμων στόχων. Ευχαριστώ πολύ Κάριν Αρνελίτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάξ που ήρθατε και που έρχεστε τόσα χρόνια εδώ και μας βοηθάτε στην επίτευξη των ε, στόχων. Όπως είπε και η Κάριν, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά κάτι γίνεται και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες έρχονται προς ε, το πλευρό μας. Ε, θέλουμε να θεωρούμαστε προοδευτική κοινωνία και δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο παρά το γεγονός ότι οι επιτροπές μας το προσπαθούν, όμως είναι μια αρχή αυτή η ομάδα. Όπως ε, και, είπε και ακούσαμε στην παρουσίαση της ε, συναδέλφου από τη Φιλανδία, χρειάζεται συνεργασία όλων έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους. Ακριβώς γιατί το θέμα αυτό είναι παγκόσμιο. Χρειάζεται φυσικά περισσότερη δουλειά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και όπως ε, έχουμε δει και στο Νταβός, η κλιματική απειλή είναι παγκόσμια. Και τις τελευταίες εβδομάδες έχω δει τεράστια κινητοποίηση από νέους ανθρώπους, βγήκαν στους δρόμους και είμαι περήφανος για αυτούς. Στην έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Εξωτερικών Υποθέσεων για την ε, περιβαλλοντική διπλωματία, για το κλίμα, έχουν γίνει πολλές καλές προτάσεις. Θέλω όμως να ρωτήσω ε, το εξή. Χρειάζεται όχι μόνο κλιματική διπλωματία, αλλά και γνώση, ενημέρωση. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διασύνδεση με την επιστήμη που αναφέρεται. Θεωρείτε λοιπόν πως Χρειάζεται διπλωματία για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης διδάσκεται αυτό το είδος διπλωματίας ε, στο πλαίσιο της εξωτερικής ε, πολιτικής, ανήκει στην εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερα τώρα που εξετάζουμε το κλίμα και το εμπόριο, ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε την σημασία και της άλλης πλευράς του Ατλαντικού με τη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες, το ρόλο της Ιαπωνίας. Πώς μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει και σε σχέση με αυτές τις εμπορικές ε, συμφωνίες έτσι ώστε να έχουμε ένα ε, στιβαρό ε, πλαίσιο και για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στον χώρο του εμπορίου. Ευχαριστώ. Ο Σαλ Γκέρντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που βλέπω τον Τζέφρι Σάξ Θυμάμαι μια φορά στο Παρίσι, στον ΟΣΑ μου είχατε πει ότι είμαι σχεδόν πάντα, κάνω σχεδόν πάντα λάθος. Ελπίζω αυτό να μην ισχύει σήμερα, αλλά από την πλευρά αυτή που ανέφερα, ήθελα να αναφέρω ανεκδοτικά το θέμα αυτό για να μιλήσω για την ουσία. Εντυπωσιάστηκα από την όλη παρουσίαση. Που... Κοιτάξτε, συμφωνούμε μαζί σας. Υπάρχει μια διακυβέρνηση ε, ανύπαρκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ε, αυτή που υπήρχε παραβιάζεται τώρα από τον πρώτο τον ΗΠΑ. Είμαστε σε κατάσταση που επικρατούσε πριν από το 1945. Ε, έχουν καταρριφθεί όλες οι πολυμερείς προσεγγίσεις. Αυτός, αυτό είναι το υπόβαθρο υπάρχει πλανητική καταστροφή. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική που μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους που παραθέσατε, βλέποντας τώρα τι γίνεται στους G7 και οι ανακοινώσει που βγαίνουν από εκεί είναι κάτι άχρωμο και άοσμο. Τίποτα δεν συμβαίνει και για τους G20 το ίδιο ισχύει. Κάναμε προσπάθειες να βάλουμε στη μερίσια διάταξη το θέμα της πρόσβασης στην κοινωνική ασφάλεια είναι στη του G20. Μα είπαν πολύ αργά αυτό να μπει στην ημερήσια διάταξη. Η αντίδραση εκείνων που δικούν τον κόσμο είναι τόσο γελία. Δεν ξέρω τι να κάνουμε, να γελάσουμε, να κλάψουμε με αυτά που βλέπουμε. Μετά υπάρχουν διάφορα βήματα συζητήσεων που γίνονται συζητήσεις, ε, προτάσεις που παραμένουν όμως σε θεωρητικό επίπεδο και, δεν, και το υπόλοιπο που υπάρχει σε επίπεδα του ε, διακυβέρνηση, που υπάρχει σε επίπεδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου τελικά και αυτό απειλείται. Λοιπόν, υπάρχουν μικροπυλώνες διακυβέρνησης παγκόσμιας. Μπορούμε να καταλήξουμε μέσω αυτών σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Δεν νομίζω για την ώρα κάνουμε βήματα οπισθοχώρησης, τουλάχιστον έτσι θα διαπιστώνω. Μια απλούστατη ερώτηση. Με εντυπωσιάζει πάντα όταν ακούω εκπροσώπους τον είπα, το ότι σκέφτονται πρώτα απ' όλα τη στρατηγική και δεύτερον δεν σκέφτονται παρά μόνο τη στρατηγική. Αν είχατε την εξουσία στα χέρια σας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήσασταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πείτε μου, πώς θα οργανώνατε το, την έξοδο από αυτό το αδιέξοδο, ε, τι αποφάσεις θα παίρνατε. Είμαστε στη χαραυγή, είμαστε εν ώψη μάλλον της, ε, των ευρωεκλογών που είναι σημαντικότατες, εξαιρετικά σημαντικές. Εάν απευθυνόσασταν ε, στην κοινή γνώμη, είχατε αυτή την εξουσία στα χέρια σας, ε, τι θα τους λέγατε. Πολύ πρωτότυπη ιδέα λοιπόν. Αναφέρουμε έναν εκπρόσωπο, τον είπα, ενώπιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω βέβαια σε ποια ομάδα θα ήσασταν οι υποψήφιες. Ο κύριος Παρνιό έχει το λόγο. Κοιτάξτε, η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που έχει την εξουσία. Εμείς το Ευρωκοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είμαστε εκλεγμένοι άμεσα αιρετοί ε, εκπρόσωποι έχουμε την εξουσία. Ε, λοιπόν, με τη σειρά μου θέλω να πω πόσο χαίρομαι που άκουσα αυτά που μας είπατε το θέμα θεωρώ ότι είναι υπόθεση του αιώνα, του 21ου αιώνα. Τώρα λοιπόν πρέπει να προετοιμαστούμε. Να προετοιμάσουμε μια κοινωνία που δεν θα χρησιμοποιεί τον άνθρακα. Αυτόν που μας παρουσιάσατε εκ νέου στην παρέμβασή σας. Και στις αρχές αυτές του 21ου αιώνα έχουμε την εντύπωση ότι περάσαμε δύσκολες στιγμές στην Κοπενχάγη το έζησε αυτό όταν ήμασταν στην ΚΟΠ όπου δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε όταν όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ήταν παρόντες παρόλα αυτά δεν ήταν ο Ντολαντρό που ήταν επικεφαλής των ΗΠΑ αλλά Μπαράκ Ομπάμα και όμως κανείς δεν κατάφερε να βρει μία λύση με την ευκαιρία αυτή της ΚΟΠ στην Κοπενχάγη. Το Δεκέμβριο του 2009, το Δεκέμβριο του 2015 ήμουν υπερήφανος για αυτή τη Συμφωνία των Παρισίων. Ήμουν εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα τον Οκτώβριο του 2015 που επέτρεψε να δείξουμε την βούληση της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εξέβρεση λύσης. Όμως αυτή η συμφωνία των Παρισιών που ήταν μια καλή ευρωπαϊκή νίκη δεν είναι περιοριστική, δεσμευτική συμφωνία. Και βλέπουμε ότι μετά το 2015 ε, έχουμε επαναχωρήσεις, οπισθοχωρήσεις. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, δεν θέλω να τα κατανομάσω, να κατανομάσω για να μην γίνομαι δυσάρεστος, αλλά κράτη-μέλη μεγάλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπαναχώρησαν. Όπως είπατε, έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ε, που είναι πιο μακροπροθέσμο. Λοιπόν, τρει μήνε πριν τι ευρωεκλογέ που θα γίνουν στι 26 Μαου, του επομένου Μαΐου, εμείς οι ευρωβουλευτέ τη επόμενη θητεία θα πρέπει να υπομισθούμε τις ευθύνε μας. Το είδαμε και στο Κατοβίτσε στην COP24. Ε, μας λείπει το θάρρος. Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν έχουμε το θάρρος. Δεν έχουμε απομειστεί τις ευθύνες μας. Ακούμε καλές ομιλίες σε κάποιες πανεπιστημιακές συναθρήσεις. Πέρα από αυτές τις ε, ομιλίες ε, θα πρέπει να μπούμε στο θέμα. Είδα Γάλλο Υπουργό δημοφιλή στη Γαλλία που παρετήθηκε διότι θεωρούσε ότι η ενεργειακή μετάβαση η οικολογική δεν προχωρούσε αρκετά γρήγορα στη Γαλλία. Αλλά ακούγοντας αυτά που μας είπατε για τον πλανήτη σε κλίμακα υπήρου ή σε κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την πολιτική που θα βαρύνει, θα επιτρέψει μάλλον θα έχει βάρος για να αλλάξουμε νοοτροπία και προσέγγιση. Συγκεκριμένη ερώτηση. Κάποιες προτάσεις που έθεσαν κάποιοι εδώ εν ώψη των ευρωεκλογών που λέει, να μπούμε στην ουσία. Ποια είναι η απόψή σας αυτό. Είμαστε σε μια φιλοευρωπαϊκή ευαισθησία που λένε ότι είναι κλιματοσκεπτικιστές οι λαϊκιστές Όπω είναι ο πρόεδρο των ΗΠΑ, που δυστυχώς δεν είναι μόνο του. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Κάνουμε προτάσεις για τη δημιουργία ενός Ταμείου Καταπολέμησης ενεργειακή Φτώχειας. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο αν θέλουμε τα λαϊκά στρώματα στην Ευρώπη να μπορέσουν να πούν ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι τιμωρία, δεν είναι κύρωση για μας αλλά το 44,5 εκατομμύρια ε, Ευρωπαίοι είναι αυτοί που έχουν ανεπαρκή πρόσβαση ε, στην ε, ενέργεια ή δεν μπορούν να έχουν το κόστος. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα του Κλίματος που θα επιτρέψει να είναι το δοχείο συλλογής όλων αυτών των πόρων που έχουμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διαθέσει, δημιουργεί ε, έχει ε, έχει δημιουργήσει ένα ποσό τεράστιο τεθεί 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη βιωσιμότητα το, του ευρώ και για να υλοποιηθούν πράσινες δραστηριότητες. Προτείνουμε να επαναπροσανατολιστούν οι προσπάθειες και οι πόροι να κινηθούν προς την οικολογική μεταμόρφωση Θέλουμε να υπάρξει και φόρος του άνθρακα που θα επιβάλλεται στα όρια, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ισχύει για τις ε, ε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν σέβονται τη Συμφωνία των Παρισίων. Τέλος, όπως είπατε, θέλουμε να βγούμε ε, από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων στην Ευρώπη. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως επιδοτούν τα ορυκτά καύσιμα 112 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο διαθέτουν για αυτό το σκοπό. Αυτή η εξάρτηση με το πετρέλαιο ε, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλη. Προτείνουμε να ξαναχρησιμοποιηθούν τα δημόσια αυτά χρήματα, διότι είναι επιδοτήσεις που δίδονται προς όφελος των ανανεωσίμων πηγών της ενέργειας και της ενεργειακής αποδόσης, κυρίως στον τομέα των μεταφορών, που είναι ένας ο τομέας που σήμερα δημιουργεί κάποιες δυσκολίες ε, στην Ευρώπη. Τέσσερις προτάσεις υπάρχουν που θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Γι' αυτό ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας επ' αυτών. Αυτές οι προτάσεις με κάνουν να λέγω ότι πρέπει να σταματήσουμε τις ε, ομιλίες, τις όμορφες ομιλίες και να υποβάλουμε και να προχωρήσουμε πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μίλησαμε λοιπόν για τις έξι πολύ σημαντικές μεταβολές ε, που προτείνεται. Θέλω λοιπόν και εγώ να ρωτήσω ποιος ο ρόλος ε, των ε, ανισοτήτων σε αυτές τις προτεραιότητες. Συμφωνώ με τα φορολογικά, όμως αναρωτιέμαι πού μπορεί να ταιριάξει το θέμα των ανισοτήτων. Σας ευχαριστώ όλους για τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Τι κάνουμε λοιπόν εν ολίγης, πού πάει ο κόσμος και πόσο δύσκολα και περίπλοκα είναι τα πράγματα. Νομίζω πως ε, θα έλεγα πως από γεωπολιτικής απόψης ε, είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να περάσει μπροστά σε διεθνές επίπεδο και να μην εξαρτάται ε, πλέον από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Να περάσει μπροστά και να αποτελέσει μια ισχυρή ε, φωνή απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, στην Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες. Διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει οτιδήποτε και να εξηγήσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση ούτε να αναλάβουν ευθύνες ούτε να ηγηθούν. Και αυτό είναι μια αλλαγή σε σχέση με τις τελευταίες δεκαετίες. Οφείλεται εν μέρη στον Τραμπ, αλλά όχι μόνο σε εκείνον. Είναι περισσότερο μακροπρόθεσμη η πρόκληση. Και προσπαθούμε στις ΗΠΑ να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω πως η πολιτική θα ανακάμψει και θα ξεπεράσει αυτή την επικίνδυνη φάση στην οποία βρίσκεται δεν νομίζω όμως ότι το συμφέρον της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου είναι το ίδιο με πριν 20 χρόνια. Δηλαδή η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Έχουμε και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η οποία επίσης πρέπει να αναλάβει ευθύνες και να γίνει σημαντικός εταίρος. Η Ευρώπη όμως δεν πρέπει πλέον να εξαρτάται από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν κοιτάζετε προ εκεί, μην κοιτάζετε, δεν θα το βρείτε κάτι τέτοιο. Μην περιμένετε από τι Ηνωμένε Πολιτείε να αναλάβουν τα ενία. Και... Ζητώ συγγνώμη που γίνομαι τόσο ευθύ, όμως το μόνο μήνυμα που έχω να δώσω για το Μάιο, για τι ευρωεκλογέ, είναι πω η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ή μάλλον ο Τραμπ προσπαθεί να υπονομεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και να προωθήσει εθνικιστικές ιδέες. Ο κύριος ε, Μπάνον, ο οποίος είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα πρόσωπα και δεν μιλάω για την εμφάνισή του αλλά για την ιδεολογία του, είναι το... Είναι η ενσάρκωση μιας ιδέας, δηλαδή ποιες ιδέες ότι ο εθνικισμός πρέπει να κυριαρχήσει, και ότι θα υπάρξει πάλι των εθνών. Είναι πολύ πρωτόγονες αυτές οι ιδέες. Η Ευρώπη τις ξεπέρασε χρόνια, δεκαετίες πριν, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει περάσει σε μία μορφή διακυβέρνησης ε, διεθνική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν λοιπόν να υπονομεύσουν αυτήν ακριβώς την διάσταση της Ευρώπης ή μάλλον η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό είναι ανόητο και πολύ επικίνδυνο. Όμως στη χώρα μου αυτούς έχουμε στην κυβέρνηση. Από τους χειρότερους που υπάρχουν. Διότι δεν μας κυβερνούν οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες, ε, οι ηγέτες, αλλά μας κυβερνούν ε, οι χειρότεροι των ε, χειροτέρων. Και δεν χρειάζεται φαντασία, ακούστε μόνο πώς μιλάει. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Η Ευρώπη όμως πρέπει να κάνει κινήσεις, να συνομιλήσει με την Κίνα. Όμως, ε, πώς θα γίνει αυτό, θα γίνει, θα γίνει 28 διαφορετικές συνομιλίες, θα γίνει ε, η συνομιλία Κίνας με 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προτιμούσε η συνομιλία να γίνει μεταξύ Ευρώπης και Κίνας και αυτό θα τέριαζε διότι υπάρχουν πολλά όμοια στοιχεία και αλληλοσυμπληρώνονται αυτές οι δύο οντότητες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μία ε, υπερεαλιστική δύναμη που πνέει τα λίστια και η Κίνα αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς είναι αναδυόμενη υπερδύναμη, θεωρείται εχθρός. Αυτό όμως είναι λάθος και πολύ επικίνδυνο σαν σκέψη και η Ευρώπη ακολουθεί αυτήν την πορεία. Να απαγορευτεί η Huawei, τα προϊόντα της Κίνας. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και παίζει η Ευρώπη με την φωτιά. Κινδυνεύει να πέσει στην ε, παγίδα της στενόμυαλης σκέψης. Και δεν νομίζω πως ζούμε ξανά το 1936, αλλά το 1910, όπου ο εθνικισμός έχει γιγαντωθεί, όπου υπάρχουν διάφορες ε, υπομάδες ε, και ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα για όλον τον κόσμο. Το μήνυμα πρέπει να είναι παγκόσμια συνεργασία έτσι ώστε να συντελεστεί αυτή η μετάβαση. Εάν εγκαταλείψουμε αυτό το όραμα τότε δεν θα καταφέρουμε τίποτα. διότι το θεματολόγιο είναι παγκόσμιο, όχι της Ευρώπης, ούτε της Γερμανίας, ούτε της Γαλλίας, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι παγκόσμιο και έχει κοινό παρονομαστή τη συνεργασία. Διαφορετικά δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα μόνοι μα, ούτε μία χώρα, ούτε μία περιφέρεια. Δεν θα καταφέρουμε να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή χωρί μία ισχυρή συνεργασία με την Κίνα. Χωρί μία συνεκτική προσέγγιση με την Ινδία. Αυτά είναι απλά μαθηματικά. Οι εκπομπές αρίων του θερμοκηπίου. Δείτε τα νούμερα. Δεν, δεν μιλάω με θεωρητικούς όρους. Για να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την ε, κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την έκκληση αερίων του θερμοκηπίου χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση και η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή, διότι αυτό είναι ζωτική σημασία και για τα συμφέροντα τη ίδια τη Ευρώπη, αλλά και για όλον τον κόσμο. Και φυσικά ξέρω πω ε, υπάρχουν προβλήματα αδράνειας, προβλήματα δομικά ε, θεωρείται πως οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι εγγυητής της ε, ασφάλειας, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αυτό που προσφέρουν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι ασφάλεια για σας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ξεκίνησαν όλους τους πολέμους στην γειτονία σας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. στη Συρία, το Ιράκ, την Λιβύη φυσικά, όχι μόνες τους, είχαν και βοήθεια. Τα έκαναν χάλια λοιπόν στην περιφέρεια της Ευρώπης, ακριβώς διότι δεν υπήρχε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική πέραν από την προειδοποίηση της Ευρώπης να μην, ε, μπει, να μην μπει η Αμερική στο Ιράκ, το οποίο ήταν πολύ ωραίο όλα, που θέλω να καταλήξω, ότι η Ευρώπη ότι η Ευρώπη χρειάζεται πέρα από την στρατηγική για τη μετάβαση και μια ε, κοινή εξωτερική πολιτική. Είναι κέρια σημασίας, διότι η Ευρώπη είναι και οι αξίες ε, τις οποίες ε, πρέπει να ακολουθούμε και να ενστερνιστούμε όλοι. Και δυστυχώς ε, πρέπει το πάθημα να μας γίνει μάθημα. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτύχει, θα αποτύχουν και όλες οι υπόλοιπες ενώσεις. ΑΣΕΑΝ, Αφρικανική Ένωση, θα αποτύχουν όλες οι προσπάθειες για περιφερειακή ολοκλήρωση. Δεν θα επιβιώσουμε από αυτόν τον αιώνα, εάν δεν αλλάξει κάτι. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, ότι ο εθνικισμός έχει οδηγήσει σε αυτά που όλοι γνωρίζετε. Αλλά η πολιτική για τη μετανάστευση, για τους ε, πρόσφυγες άλλαξαν, αναποδογύρισαν την πολιτική της Ευρώπης και οι Ηνωμένε Πολιτείε χρειάζεται να σταματήσουν όλους αυτούς ε, τους ε, πολέμους ε, που διεξάγουν, να σταματήσουν την κλιματική αλλαγή για να σταματήσουν και οι προσφυγικές ροές. Η Ευρώπη σχεδόν κατέρευσε με το προσφυγικό. Και το προσφυγικό ήταν αυτό που επικράτησε εις βάρος όλων των ε, υπόλοιπων θεμάτων. Όμως αυτό δεν πρέπει να είναι το κεντρικό κομμάτι της πολιτικής σας. Η κεντρική πολιτική πρέπει να είναι η παροχή αξιοπρεπούς ε, διαβίωσης, βιώσιμης ανάπτυξης σε έναν ενωμένο ευρωπαϊκό χώρο με μια ισχυρή ασφάλεια την οποία θα είστε σε θέση μόνοι σας να παρέχετε ε, και να συνεργάζεστε με τις γειτονικέ ε, και μη περιοχές, με την Κίνα, με την Νοτιοανατολική Ασία, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Αφρική, ως μια ισχυρή ενωμένη φωνή. Και με τη σημερινή της μορφή, η ηγεσία των ε, Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ δυσκύλια, προσπαθεί να υπονομεύσει αυτή τη συνεργασία μέρα με τη μέρα, βήμα-βήμα. Ακόμα και ο πρόεδρος Ομπάμα, ο οποίος ήταν αξιόλογος, δεν ήταν αρκετός, διότι είναι μόνο ένα. Η Ευρώπη πρέπει να δουλέψει περισσότερο από ποτέ, διότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε εποχές ψυχρού πολέμου όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν ο εγγύτης της ε, ασφάλειας. Πρώτα λοιπόν πρέπει να λύσετε τα της ασφάλειας εντός Ευρωπαϊκή Ένωσης έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ισχύρη Ενωμένη Ευρώπη που θα μπορέσει να γυθεί και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω πως το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Αλλά γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Κίνα εχθρό. Πρέπει να καταλάβετε την ιδεολογία των ΗΠΑ, η οποία φαίνεται σε κάθε πτυχή της πολιτικής, σε κάθε έγγραφο. Και αυτή είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι η ισχυρότερη δύναμη. Τελεία. Αυτή είναι η ιδεολογία των ΗΠΑ οι Ηνωμένε Πολιτείε πρώτες, δυνατότερες. Αυτό βέβαια δεν είναι βιώσιμο για να εγγυηθεί την ειρήνη στον κόσμο. Είναι μια ιδεολογία πάρα πολύ επικίνδυνη και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Και πρόβλημα μάλιστα που σας αφορά, διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε όταν βλέπουν την επιτυχία οπουδήποτε αλλού εκτός από το εσωτερικό τους, τη θεωρούν απειλή, διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θέλουν ίσους επιτυχημένου Ετερούς θέλουν κυριαρχία, πρωτοκαθεδρία. Για αυτό προβλέπει και η εθνική στρατηγική, τον είπα, για την ασφάλεια. Primacy, αυτή είναι η λέξη παντού. Η Κίνα είναι εχθρός, η Κίνα δεν γίνεται όμως να είναι εχθρός ε, της Ευρώπης, ε, διότι είστε στην ίδια ήπειρο, δεν σα χωρίζουν ωκεανοί. Χρειάζεται τα προβλήματα να λυθούν ειρηνικά και με τρόπο συνεργατικό, με διασυνδεσιμότητα. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές ε, για να μην είμαι τόσο αόριστος και μιλώ αφηρημένα. Ελπίζω λοιπόν η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε ένα χρόνο να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τους παρουσιάσει συγκεκριμένε, κατευθυντήσαμε συγκεκριμένου συγκεκριμένους οδικούς χάρτες για την αλλαγή της χρήσης ε, τη γη, για τη βιώσιμη ε, ενέργεια και ανάπτυξη και για όλους τους υπόλοιπου τομείς ε, στου οποίους χρειάζεται αλλαγή. Να μην ε, μιλά γενικά, να μην μιλάμε και να αναφέρεται σε στόχους, σε οδικούς χάρτες. Μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε συγκεκριμένη πρόταση μπροστά μας. Φυσικά οι επιμέρους χώρες θα έχουν τις δικές τους εθνικές πολιτικές. Όμως χρειάζεται η δημιουργία ενός πλαισίου σαφούς και κατανοητού. Διότι σε πολλούς τομείς ε, της ε, ζωής μας δεν περιμένουμε συντονισμένη πολιτική, δεν περιμένουμε ας πούμε ε, την κάθε χώρα να δημιουργήσει δική της πολιτική για το 4G, για το 5G, για το διαδίκτυο, ή για, την, για, τους, ανα, τους ε, ελέγχους κυκλοφορίας. Αυτά είναι πρότυπα τα οποία θεσπίζονται είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε περιφερειακό. Γι' αυτό λοιπόν ε, παρομοίως και για την ενέργεια και για τις μεταφορές και για να σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ σύντομα θα πω ότι η οικονομία της Ευρώπης στηρίζεται αναμφίβολα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο τομέας αυτός σε 15 χρόνια θα είναι τελείως διαφορετικός. Θα αλλάξει 100% θα γίνει ηλεκτρικός, ε, θα υπάρχει περισσότερη αυτονομία, θα υπάρχει περισσότερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καμία σχέση με τα 100 τελευταία χρόνια. Η επιτυχία λοιπόν της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας εξαρτάται από αυτήν την ικανότητα και την ταχύτητα της μετάβασης. Διαφορετικά όλοι θα οδηγούμε κινέζικα αυτοκίνητα και θα οδηγηθούμε σε περιβαλλοντική καταστροφή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν χρειάζεται δουλειά, χρειάζονται προγράμματα τα οποία να συμβαδίζουν με τις ε, εξελίξεις και τις αλλαγές. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα έλεγα πως όχι. Λέμε πως μέχρι το 2030 τα οχήματα που θα πολλούνται θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών. Τι εννοείται με αυτό. Γίνεται πιο σαφής. Φτιάξτε υποδομές για οχήματα ε, που χρησιμοποιούν υδρογόνο ή ηλεκτρισμό, δώστε να καταλάβουν οι υπόλοιπε χώρε τι πρέπει να κάνουν και παράσχεται την κατάλληλη υποδομή, έτσι ώστε και οι οδηγοί να ξέρουν πως ε, τα οχήματα που θα οδηγήσουν θα είναι ακόμα καλύτερα από αυτά που παράγονται τώρα. Και σίγουρα τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, όμως όταν θα είναι πιο έξυπνα, όταν θα χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια θα είναι ακόμα καλύτερα. Και έτσι θα συντελεστεί η μετάβαση, η αλλαγή αυτή στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν σας ε, παροτρύνω να πιέσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει οδικούς χάρτες. Να εξηγήσει στους ηγέτες ε, στο Συμβούλιο ότι αυτή η αλλαγή δεν θα γίνει μεμονωμένα, ακόμα και αν ορισμένοι θεωρούν πως ε, το πολιτικό τους ε, μέλλον εξαρτάται από την έμφαση στα εθνικά ζητήματα, να τους δώσετε να καταλάβουν ότι δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να περάσει σε αυτή τη νέα εποχή. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα που θα ήθελα να τονίσω και το κύριο μήνυμα που θέλω να δώσω. Σίγουρα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό το σκεπτικό και στην εμπορική πολιτική. Χρειάζεται αναθεώρηση, διόρθωση της φορολογικής πολιτικής ε, εάν κάποια χώρα δεν ε, συμμορφώνεται με την νομοθεσία για την αποδέσμευση από άνθρακα. Όμως πιστεύω πως είναι εφικτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αλυσίδες αξίας δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Θα έλεγα όμως ότι χρειάζεται να εντοπιστούν οι κυριότεροι τομείς όπου παρατηρούνται δυσκολίες στις αλυσίδες αξία, Δηλαδή, σε γενικέ γραμμές, ο καφές, το φινικέλαιο, η γεωργία, ε, η σόγια, η εξορυκτική βιομηχανία, τα ορυκτά καύσιμα και οι τομεί όπου δραστηριοποιούνται ε, όπως η κλωστοϊφαντουργία ας πούμε σε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ε, βαριά εργασία. Χρειάζεται λοιπόν να ζητήσουμε τη γνώμη των ε, διαφορών ε, βιομηχανικών ενώσεων ή ενώσεων ε, παραγωγών έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα, την παιδική εργασία, την καταναγκαστική εργασία, την ρήπανση, τη μόλυνση, αποψήλωση των δασών κτλ. Μετά περνάμε σε άλλο στάδιο, στην υποβολή εκθέσεων. Και εδώ κάθε κρίκος της αλυσίδας αξίας πρέπει να υποβάλει εκθέσεις, πρέπει να ε, του ασκείται έλεγχος των αποτελεσμάτων ε, για να καταφέρουμε να αξιολογήσουμε το, προ, το μέγεθος του προβλήματος. Και μετά θα επέβαλε οικονομικές κυρώσεις σε μια περίοδο τριετή, πενταετή, αν αποδειχθεί ότι γίνονται εισαγωγές από έναν προμηθευτή ο οποίος καταφανώς έχει παραβεί τις προδιαγραφές της αλυσίδα αξιών όσον αφορά την εργασία παιδιών ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά. Εγώ θα επέβαλα οικονομικές κυρώσεις ξεκινώντας με περιοχές που ε, είναι επικίνδυνες, έλεγχο και απαιτήσει για υποβολή αναφορών και εκθέσεων και με ισχυρότατο ρόλο των συνδέσμων των βιομηχανικών εντός των διαφόρων τομέων. Διότι όλοι αυτοί οι τομείς έχουν τους δικούς τους φορείς. Ο τομέας του καφέ έχει την παγκόσμια πλατφόρμα του καφέ και ο κάθε τομέας έχει την πλατφόρμα του. Εγώ θα τους έβαζα να αντιμετωπίσουν ε, οικονομικές κυρώσεις αν δεν συμμορφωθούν με κοινωνικές προδιαγραφές, προδιαγραφές για την εργασία και για το περιβάλλον. Είναι κάτι εφικτό πιστεύω. Αυτό θα βοηθούσε και τους διάφορους τομείς στο εσωτερικό να επιβάλλουν τη σωστή συμπεριφορά στα μέλη τους παρά να κινούνται ανεξέλεγκτα που αυτό είναι κάτι που δημιουργεί δυσκολίες. Στο θέμα των ανισοτήτων τεχνικά είναι στην πρώτη μεταμόρφωση. Έχουμε τη μεταμόρφωση που αποτελείται δεξιότητα, απασχόληση, παιδεία ε, και ανισότητες. Εκεί ανήκει αυτό το θέμα. Αλλά και η Ευρώπη είναι η πιο κατάλληλη περιοχή στον κόσμο για τη μείωση των ισοτήτων. Ε, λοιπόν, συστηματικά διάφοροι συντελεστές του, είναι κάτω από άλλες περιοχές του κόσμου στον αφορά την κοινωνικό αποκλεισμό. Είσαστε σοσιαλδημοκρατικό ε, μοντέλο που ενέπνευσε ε, την πολιτική στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι κάτι που συνεχίζεται μέχρι τώρα. Λοιπόν, εγώ θα έβλεπα τους διάφορους δείκτες ε, του, εθνικού εισοδήματος. Είναι οι, μόνοι, είναι οι βορειοευρωπαϊκές χώρες έχουν ε, κάτω από 0,3. Οι διαφορές μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης είναι πολλές, αλλά μία από τις διαφορές είναι ότι η Ευρώπη επιβάλλει αρκετούς φόρους και κατανέμει τους πόρους για να ελέγχει τις ανισότητες. Και αυτή είναι η ουσία της επιτυχίας, διότι οι δυνάμεις της αγοράς μας ε, είναι φυγοκεντρικές. Χρειάζονται φορολογικές κεντρομόλε δυνάμεις και αυτό είναι ο πυρήνα για μείωση των ισοτήτων πέρα από τι αξίε των ανθρωπινών δικαιωμάτων, ισότητα των φύλων κλπ. Είναι το σύστημα φορολογικών μεταφορών, μεταφορά και διανομή των πόρων που βοηθά να μειωθούν οι ανισότητε. Ε, ή να υπάρχουν συνδικάτα, δυνατότητε συναπόφαση κλπ. ώστε οι εργάτε συμμετέχουν και επιχειρήσει να μην κινούνται ανεξέλεγκτε και να προωθούν εσωτερικά τι ε, διάφορε ανισότητε στι χώρε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον ομιλητή μας. Χειροκοτώντας τον και μας υπενθύμησε ότι κινούμεθα προς τις καθοδόν εκλογές που μας υπενθύμησε τη σημασία που έχουν αυτές οι εκλογές και όπως είπε οι σημασίες του είναι, η σημασία του είναι ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. λέω Βρετανίδα και βλέπω συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι εδώ. Εμείς χάσαμε με, μετά την επίθεση ε, όπως, ανθρώπων όπως τον Μπάνον στο Ηνωμένο Βασίλειο χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Ε, την, ε, το πιστεύω μας για την Ευρώπη και να υποστηρίξουμε την Ευρώπη. Δεν έπρεπε να απολογούμεθα για το έργο που κάνει η Ευρώπη. Και το μήνυμα πάνε στις εκλογές είναι να είναι ισχυρό το μήνυμα. Αυτό που συμβαίνει εδώ έχει σημασία, πρέπει να το δείξουμε. Και μεταμορφώνει τον υπόλοιπο κόσμο αυτό που γίνεται εδώ. Και μπορεί να γίνει καλύτερο ο κόσμο και καλύτερη ζωή των ανθρώπων που εκπροσωπούμε και καλύτερη ζωή για όλου του ανθρώπου στον κόσμο. Αν η Ευρώπη πετύχει σωστέ λύσει, αυτό θα είναι ένα ισχυρότατο μήνυμα για την υπόλοιπη υφήλιο. Και αυτό είναι θετικότατο μήνυμα από την πρωινή συζήτηση και αυτό να πάρουν μαζί του οι συνάδελφοι. Συνάδελφοι, ευχαριστούμε τον Τζέφρι. Ολοκληρώθηκε η ακρόση. Ακούσαμε τον κύριο Τίμερμαντς και τον Τζέφρι Σάξ και πάμε στο σημείο 4 της κοινή μας συνεδριάσεως μεταξύ Επιτροπής Περιβάλλοντος και Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα εξετάσουμε την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που συνετάχθη γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι πριν από τις εκλογές. Έχουμε το έγγραφο προβληματισμού που κατέφθασε τώρα. Έχουμε πάρει από την διάσκεψη των Προέδρων και των Προέδρων Επιτροπών για τη σύνταξη μια εκθέσεω πρωτοβουλία, ούτω ώστε να συμβάλλει το Κοινοβούλιο μέσω του κειμένου στην προετοιμασία του πολιτικού φόρουμ του Σεπτεμβρίου του ΟΗΕ και υπάρχει στο ΣΥΜΠΙΟΥ τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής και θέλαμε να συμβάλλει σε εργασίες του Συνόδου Κορυφής στο Κοινοβούλιο. Ο Ζιλ Παγνιό θα πάρει το λόγο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα προεδρεύσει τι συζητήσει αυτή. Ζήλε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Λίντα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές των δύο επιτροπών για την πολύ καλή συνεργασία που ε, έτσι θέσαμε ένα πλαίσιο εργασιών ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς συνεργασία αυτή δεν θα ήταν ε, δυνατόν. Όπως είπε η Λίντα Μακέβαν, λοιπόν έχουμε αυτή την έκθεση της στρατηγική και συμμετοχή στο βήμα αυτό των συζητήσεων. Οπότε θα θέσουμε στο επίκεντρο του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, στο επίκεντρο των εργασιών του Κοινοβουλίου για πολλά έτη. Έχουμε πολύ ψωμί να φάμε ακόμα για να πετύχουμε του στόχου του θεματολογίου του 2030, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημαντική εργασία που έγινε για να ε, μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τι διεθνεί υποχρεώσει μέσω των πολιτικών σοφορά το θεματολόγιο του 2030 ή τη Συμφωνία των Παρισίων του Δεκεμβρίου του 2015. Η δράση για το κλίμα, όπω γνωρίζετε, είναι ένα από του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη που εξετάστηκε ει βάθο φέτο στο, στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου σε σχέση με του αναθεωρημένου στόχου φέτο και το γενικό θέμα του Φόρουμ ε, του 2009 που είναι αυτονομία των ανθρώπων και να εξασφαλίζεται η ισότητα, των ισοτήτων. Αυτά είναι θεμελιώδη θέματα. Θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές, Φανσές Καμπούς και την κυρία Ελένη Θεοχάρους, για τη συνεργασία τους. Έχουμε τώρα ένα 20 λεπτό για την παρουσίαση και συζήτηση του σχεδίου εκθέσεως. Καθυστερήσαμε λίγο, θα δώσω το λόγο σε εκείνο που αντικαθιστά τους συνεισηγητές που δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ σήμερα. Ο για τον κύριο Γκαμπής Δίνω το λόγο στον κύριο Σόνικ, ο οποίος είναι εδώ να εκπροσωπήσει τον κύριο Γκαμπίους. Έχετε το λόγο. από πλευρά του κυρίου Γκάμπου, που δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί <clears throat> θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά σχόλια που προετοίμασε ο εισηγητή από πλευρά ΣΕΛΚ, ο κύριος Γκάμπου. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Γκάμπου πιστεύει ότι η δράση της Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του θεματολογίου του 2030 πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι μόνο από πλευρά ευρωπαϊκή, αλλά λαμβάνοντα υπόψη και το ρόλο πρωτοπορία που έχουμε. Πρέπει να συνεργαστούμε με άλλε χώρε και πρέπει να ενθαρρύνουμε την Κίνα και τι ΗΠΑ να παίξουν ενεργό ρόλο. Ως παγκόσμια πρωτοπορία πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά επίσης πρέπει να έχουμε και κριτική σκέψη. Ο συνεισηγητής χαιρετίζει το έγγραφο προβληματισμού που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θεματολόγιο του 2030 συνδέεται με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τις συνθήκες. Πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε την πολιτική μας και να επιτύχουμε τους στόχους. Τώρα η έκθεση αυτή καθε αυτή είναι η πρώτη από μια ολόκληρη σειρά εκθέσεων που θα κάνουμε για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Το κείμενο είναι γενικόλογο και εστιάζει επί των στόχων που θα πρέπει να αναθεωρηθούν το 2019 εκπαίδευση, αξιοπρεπής εργασία, ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων, κλιματική αλλαγή, ισχυροί θεσμοί και ε, εταιρικές σχέσεις, συνεργασίες. Ο εισηγητής ε, έχει υπόψη του ότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί στόχοι που έχουν να κάνουν με την υγεία, την επιστηστική ασφάλεια και την οικονομία. Αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε στους ε, προηγούμενους εν ώψη της ε, συζήτησης και του φόρουμ υψηλού επίπεδου που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Κάθε χρόνο θα πρέπει να καθορίζουμε κάποιες προτεραιότητες <clears throat> ανάλογα με τη στιγμή στον κύκλο ε, προώθησης γιατί αλλιώ θα λέμε τα ίδια κάθε χρόνο. Τώρα, η εθελούσια εθνική αναθεώρηση. Ο εισηγητής ενθαρρύνει τα, τα κράτη-μέλη να κάνουν συνολικές και συστηματικές ε, διάμεσες αναθεωρήσεις. Και οι δράσεις μας πρέπει να είναι συγκεκριμένες μετά από τις αναθεωρήσεις αυτές. Κάποια κράτη-μέλη καλούνται από την έκθεση να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα εθελούσιας εθνικής αναθεώρησης. Γιατί δεν το κάνουν όλα τα κράτη-μέλη. Το θεματολόγιο του 2030 πρέπει να γίνει σεβαστό και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει σφαιρική προσέγγιση. Όλοι οι συμβαλόμενοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συμμετάσχουν και το σύστημα θα έχει πολλαπλά επίπεδα. Η φωνή της Ένωσης πρέπει να εισακουστεί. Η κλιματική διπλωματία μας πρέπει να ενισχυθεί. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και από κοινωνική και περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση. Ο συνεισηγητής ελπίζει να υπάρξει ομαλή συνεργασία με τον άλλο συνεισηγητή, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά χρειαζόμαστε ένα καλό κείμενο και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει πολύ καλή πολιτική βούληση από πλευρά Σόνικ και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόνικ για την ε, παρουσίαση των απόψεων του κυρίου Κάμπου. Κανεί δεν αντικαθιστά την κυρία Θεοχάρους, οπότε θα δώσω το λόγο τώρα στους Κιώδης. Κύριε Σόνικ, θέλετε να μιλήσετε και πάλι ω κοιόδη εκ μέρου σα προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο συνσηγητές. Είναι πολύ καλό έγγραφο. Σημερίζομαι τις απόψεις που εκφράστηκαν Οι στόχοι που θα εξεταστούν προσεκτικά τον Ιούλιο στην πλατφόρμα των ε, Ηνωμένων Εθνών πρέπει να είναι ε, οι στόχοι που θα μας απασχολήσουν και μας. Έτσι θα συμβάλλουμε σε αυτήν τη συζήτηση που θα γίνει λοιπόν αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται των ε, δράσεων για να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και για να είναι οι στόχοι αυτοί συνδυασμένοι με άλλους ε, διεθνείς στόχους για την ανάπτυξη των, ε, για την ε, εκπόνηση καλύτερα δικτών και για τη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κάποια κράτη-μέλη κάνουν εθελούσιες αναθεωρήσεις των βιώσιμων στόχων. Οι τροπολογίες μου θα αναφερθούν φυσικά στο θεματολόγιο 2030 και θα ασχοληθούν ακριβώς με τους στόχους που θα αναλύσουμε λοιπόν τον προσεχή Ιούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόνικ. Και τώρα οι υπόλοιποι σκιώδες. Κάντενμπαχ και μετά Γκέρεντς. Κάριν. Ευχαριστώ πολύ γενικά για την κατεύθυνση αυτής μας της ε, κοινή συνεδρίασης γιατί νομίζω ότι έτσι ε, επιβεβαιώνεται η ουσιώδη σημασία επίτευξη αυτών των στόχων. Και το μήνυμα δεν πρέπει να περιοριστεί ε, μεταξύ των μελών ΝΤΕΒΕ και ΕΝΒΗ, πρέπει να περάσει και στις άλλες επιτροπές και συναδέλφους. Ευχαριστώ για την εκπόνηση αυτής της ε, ήδη πολύ καλής έκθεσης από τους δύο συνσηγητές. Ξέρω ότι επειδή περιοριζόμαστε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα όσα θα θέλαμε και που είχαμε συμπεριλάβει αλλά πρέπει να κάνω κάποιες ε, διορθώσεις. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνοχή μεταξύ των στόχων και της χρηματοδότησης. Δηλαδή, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι για την επίτευξη των στόχων αυτών και αυτό ισχύει και για τις ε, μεσοπρόθεσμες, μάλλον τις ε, πολυετής πολυετής καλύτερα, δημοσιονομικές προοπτικές. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα πώς αξιοποιούμε τις πιστώσεις για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Επίσης, είναι πολύ πλήρης αυτή η έκθεση και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να μπει παντού σε λεπτομέρειες να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένα. Στην καταπολέμηση του ιού της ε, υπατήτηδος. Θα το αναφέρω αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό σχετίζεται με τις περαιτέρω βελτιώσεις της πρόσβασης στην υγεία και για να υπάρξει ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη στον τομέα αυτό. Ξέρω ότι με αυτό συμφωνεί και ο συνάδελφος Μποζόη και ναι μεν είναι λεπτομεριακό αυτό το θέμα αλλά ελπίζω να υπάρξει στήριξη από πλευράς των συναδέλφων και ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσω τον συνάδελφο που είναι εδώ δίπλα μου, τον Σεμ Ντάντς ο οποίος με βοήθησε, ήταν ο συγγητή πέρυσι και με βοήθησε πολύ στην, ε, ε, στο καθορισμό της θέση μου. Ευχαριστώ και τώρα ο Σαρλ Γκέρεντ. Ευχαριστώ. Ε, Έχοντα ακούσει τον Τζέφρι Σάξ, είναι δύσκολο να βρει κάτι πρωτότυπο να πει κανεί για τα θέματα αυτά. Αλλά να μιλήσω για τη χρηματοδότηση των στόχων αυτών. Πρώτα απ' όλα για την ε, δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη. Εδώ και χρόνια θέλουμε να υπάρχει μια επιτήρηση της χρήσης της. Πώς την ε, ε, διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη αυτές τις προσπάθειες. Όλοι λένε ότι πρέπει να ε, βοηθήσουμε και να είμαστε γενναιόδοροι, αλλά όταν ε, τίθεται το θέμα να βάλει κανείς το χέρι στην τσέπη, είναι πολύ πιο διστακτική. Θα επανεποβάλλω λοιπόν μια τροπολογία για την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Συγγνώμη που την επανυποβάλλω, αλλά δεν ελήφθη υπόψη. Από το Κοινοβούλιο βεβαίω, αλλά η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει οπωσδήποτε να δεσμευτούν για την τήρηση αυτών των στόχων. Δεν κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απαιτήσουν από τα κράτη-μέλη να έρθουν να λογοδοτήσουν και στα εθνικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πόσα δίνουν. Κάτι ακόμη. Συζητούμε το NDICI. Και το θέμα είναι αν πρέπει να μείνουμε στο 25% για τη χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής να πάμε στο 30% ή παραπάνω. Αυτό το θέμα πιστεύω ότι είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με το πώς <clears throat> τα κράτη-μέλη και γενικά η διεθνής κοινότητα θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη κινητοποίηση <clears throat> των 100 δισεκατομμυρίων ετησίως που χρειαζόμαστε για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Ακόμη περιμένω να δω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Ποιο θα δώσει τι. Ό,τι μπορεί να μετρηθεί πρέπει να μετρηθεί, να δοθεί ως αριθμητικό στοιχείο. Και θα πρέπει να μας πει και το Βατικανό να μας πει τι γίνεται. Όλες αυτές οι πλευρές συνδέονται. Αν δεν προσέξουμε, η χρηματοδότηση για την οποία όλοι δεσμεύθηκαν στο Κατόβιτσε, που ήταν επανάληψη μιας άλλης ε, υπόσχεσης που είχε γίνει στο Παρίσι. Εάν δεν γίνει πραγματικότητα αυτή η υπόσχεση, τότε θα ζητηθεί από τον ενωσιακό προπολογισμό να εξευρεθούν πόροι για θέματα, για το θέμα δηλαδή της ε, κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα τα πάρουμε από την καταπολέμηση της φτώχειας. Δεν είναι δυνατόν ε, ε, να μην κάνουμε και τα δύο αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια κάποια λογική και συνέπεια και καλή βούληση. Και να γίνει να γίνουν σεβαστά και τα κοινοβούλια, να έρθουν να λογοδοτήσουν. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ξεφτελιζόμαστε με αυτά που κάνουμε. Λέμε αυτά που κάνουμε, είμαστε φιλόδοξοι, λέμε τι θα κάνει η Ευρώπη και αυτό το μικρό εμπόδιο δεν μπορούμε να το υπερβούμε. Ευχαριστώ Σάρ για την παρέμβασή σας. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Όχι. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον Κασπά Φοντινή που είναι τμήματάρχη στη Γενική Διεύθυνση Ντεύκο για να μας δώσει την άποψή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να σχολιάσω την εξωτερική διάσταση της έκθεσης. Μετά θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Άστριτ Σούμαχα για να σχολιάσει τα θέματα εφαρμογής σε εσωτερικό επίπεδο. Εξωτερικές πτυχές. Πάμπολα στοιχεία της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου θεωρούμε ότι είναι πολύτιμα. Τα εκτιμούμε οι εξωτερικές και εσωτερικές πτυχές να λαμβάνονται υπόψη συνολικά. Και όπως αναφέρθηκε θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρέπει και διεθνώς να δίνει το παράδειγμα. Δεν θα εφαρμοστεί αυτό το θεματολόγιο αν δεν συμφωνούν όλοι. Επίσης, θετικότατο το ότι έκθεση σωστά τονίζει ότι η εφαρμογή και η υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι προς όφελος και της Ευρώπης όχι μόνο για άλλε αναπτυσσόμενες περιοχές, αλλά και για την Ευρώπη, σωστά αναφέρεται η ανάγκη κινητοποίηση όλων των μέσων εφαρμογής. Όπως είπε και ο κύριος Γκέριντ, ανελήφθη υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσουμε το 0,7 και 0,6 για τους στόχους αυτούς και να κινητοποιήσουμε και άλλους πόρους, ιδιωτική χρηματοδότηση, εσωτερικούς πόρους, και όλες τις αναγκαίες πολιτικές, πέρα από τα ποσοστά του ΑΕΠ. Αρκετά χρήσιμο ήταν να αφαιρθεί και υποστήριξη που να δώσουμε σε διάφορες χώρες να ενστερνιστούν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αναφέρομαι κυρίως στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες και όχι μόνο αυτό. Εκτιμούμε και τη σαφή αναφορά τη συνθήκη που επιβάλλει την υποχρέωση να λάβουμε υπόψη την αναπτυξιακή συνεργασία σε άλλους Τομεί που επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι θέμα συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, βασικό στοιχείο υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Σχετικά με αυτό, να σας πω ότι δημοσιεύσαμε την έκθεσή μας όσον αφορά το θέμα αυτό, μαζί με το έγγραφο προβληματισμού. Ενδιαφέρον άγνωσμα. Θέλουμε να αναφέρουμε το, το μείγμα εξωτερικής εφαρμογής και εσωτερικής εφαρμογής των στόχων. Και αυτό το σημείο διαπαφής θέλουμε να τονιστεί στην έκθεση. Τέλος, η έκθεσή σας σωστά αναφέρει το θέμα υλοποιήσεως των στόχων αναπτυξιακής συνεργασίας μέσω των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας. Μαζί με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους εμπλεκομένους φορείς θέλουμε να προχωρήσουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω την έκθεση. Ελπίζουμε να εγκριθεί τον Απρίλιο. Θα λάβουμε υπόψη τα βασικά μηνύματα της εκθέσεώς σας στην έκθεση αυτή. Στόχος είναι να υποβληθεί τον Ιούλιο, να παρουσιαστεί τον Ιούλιο ε, στη Νέα Υόρκη στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου. Ίσως θα ήταν χρήσιμο τώρα να αναφερθώ σε κάποιο θέμα πέρα από αυτά που μας αρέσουν, ένα θέμα που θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω. Συγγνώμη Κασπάρη, υπάρχουν πολλοί που μιλάνε, γίνεται λίγη φασαρία. Ξέρω θα ξεκινήσει η ψηφοφορία στην ΤΕΒΕ, παρακαλώ λίγη ησυχία. Θα πει σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να τα ακούσουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να αναφέρω, κάτι που αναφέρθηκε επανειλημμένα σήμερα, η έκθεση θα μπορούσε να τονίσει το όφελος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν διεθνώς στο θεματολόγιο. Αναφέρεται στην έκθεση, όπως έδειξε όμως και η συζήτηση, ίσως είναι μια πτυχή που θα μπορούσε να απτυχθεί περισσότερο. Το ίδιο να πω ότι το θεματολόγιο αυτό ε, γιατί υποστηρίζει τον, την πολυμερή προσέγγιση πέρα από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Το αναφέρει κάπως η έκθεση αλλά είναι μια σημαντική πτυχή που ίσως θα έπρεπε να τονιστεί περαιτέρω. Αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και αυτό. Η συνένεση αυτή για την ανάπτυξη ευρωπαϊκή είναι ένα εργαλείο για να διαθώσουμε την αναπτυξιακή πολιτική η οποία θα βοηθήσει άλλες χώρες να εφαρμόσουν το θεματολόγιο του, 20, του 2030 και να γίνει βιώσιμο το θεματολόγιο του 2030 θα είναι βιώσιμο εάν εφαρμόσουν την προσέγγιση αυτή όλες οι χώρες του πλανήτη. Θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω πολιτικού διαλόγου και μέσω των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να αναφέρεται εκτενέστερα στην έκθεση. και η αναγκαία υποστήριξη για τις εθνικές αιτήσιες αναθεωρήσεις και επισκοπήσεις σε τρίτες χώρες. Και αυτό μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να αναφέρω δύο πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να αναφέρονται. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων και το άλλο η νέα εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ μετά την ε, Συμφωνία του Κοτονού είναι σημαντικότατη μοχλή που θα μας βοηθούσαν να προωθήσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε εξωτερικό επίπεδο. Και θα πρέπει στις συζητήσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και τα νέα μέσα θα πρέπει να συζητήσουμε την ανάγκη υποστήριξης της υλοποίησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά είναι τα σχόλια σε αυτή τη φάση. Βέβαια είμαστε στη διάθεσή σας να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σωμάχη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συνεκτική πολιτική βλέπετε πως ε, φαίνεται και από εμάς Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη και Περιβάλλοντος. Θα συνεχίσω λοιπόν ε, στο ίδιο ύφο με τον ε, συνάδελφο. Θα σας ε, προσκαλέσω να διαβάσετε το έγγραφο προβληματισμού και θα δείτε όταν το κάνετε πώς αναφέρονται πολύ σημαντικά θέματα τα οποία βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακριβώς όπως και στην Επιτροπή σας. Δηλαδή η στρατηγική δράση βασισμένη στη συνεργασία και να είμαι πιο συγκεκριμένη. Ο πρώτος αντιπρόεδρο το είπε και σήμερα το πρωί, Καλωσορίζουμε ορίζουμε την ε, συνεργατική πολιτική βασμένη συνεργασία. Η έκθεση για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μας έδειξε πόσο σημαντικό είναι αυτό και υπάρχει εκτός από την πλατφόρμα και υπάρχουν και άλλα μοντέλα κυκλικής ε, οικονομίας για παράδειγμα που δεν θα έφταναν σε τέτοια σημεία επιτυχίας εάν δεν είχαμε υιοθετήσει τέτοια συμμετοχική προσέγγιση. Επίσης, ε, συμφωνούμε και εμείς μαζί σας για τη σημασία του ελέγχου. Ο έλεγχος εξυπακούεται πώς ε, πρέπει να γίνεται. Να σας υπενθυμίσουμε και τις ε, μελέτες που έχουν γίνει για το περιβάλλον και για τους σχετικούς δείκτες, οι οποίοι θα παρουσιαστούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος τη συνέχεια του 2019. Μετά είναι πολύ σημαντική η συνεκτική πολιτική και το mainstreaming στις, ε, στο σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Φυσικά παραμένουν προκλήσεις ε, σε θέματα εσωτερικής πολιτικής. Εδώ χρειάζεται να καταβάλουμε προσπάθειες για να γίνουν πιο συνεκτικά. Βέβαια, η Κομισιόν έχει σημειώσει πρόοδο στο εσωτερικό της, όμως όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς, ε, υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Τονίσατε και εσείς ε, πόσο σημαντική είναι καλύτερη η νομοθεσία για την επίτευξη της ε, συνοχής, για να θωρακιστούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και στην ανακοίνωση του 2016 τονίζουμε το ίδιο θέμα. Πιστεύουμε πως χρειάζεται σταδιακά να βελτιωθεί ε, η πολιτική μας ε, μέσω της ε, σύστασης ενός ανεξάρτητου συμβουλίου που θα ελέγχει την πολιτική. Σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να μειωθούν τα εμπόδια και το κενό ανάμεσα στην κοινωνική πολιτική και στην οικονομική πολιτική. Φυσικά μπορούν να γίνουν πολλά ακόμα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να γίνει κάποιο τεστ βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές. Υπάρχουν πολλές ιδέες, τις εξετάζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναπτύσσουμε πολλά σενάρια, ιδιαίτερα το σενάριο 1 που σας παρουσίασε ο Πρόεδρος Τίμερμαν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας, απόψε σας. Κύριε Σόνικ, θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση ή δεν χρειάζεται. Όχι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μέσω της ενεργού συμμετοχής τους υπογραμμίζουν το θεμελιώδη ρόλο των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σημαντική σχέση που υπάρχει μεταξύ της υλοποίηση του θεματολογίου 2030 και της Συμφωνίας των Παρισίων του Δεκεμβρίου 2015. Εύχομαι στους συνεισηγητές και σκιώδεις ε, καρποφόρες συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, ούτως ώστε να καταλήξουν σε μια, σε μια ισχυρή και φιλόδοξη θέση του Κοινοβουλίου. Και να δώσω το λόγο στην Λίντα Μακάβεν για την, ε, τα δικά της πορίσματα και το περαιτέρω χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ συνάδελφε. Το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες είναι πολύ σφιχτό. Αύριο το πρωί 10 η ώρα και μόνο αγγλικά. Γιατί έχουμε πιέσει λόγω τέλου τη θητεία. Την έκθεση την έχετε λάβει εδώ και κάποια εβδομάδα, κα, καμιά εβδομάδα. Οπότε νομίζω ότι είχατε χρόνο. Θέλω παρακαλώ να σας πω δεν υπάρχει καμία περαιτέρω δυνατότητα αναβολής. Αύριο 10 ώρα το πρωί. Για τις τροπολογίες. Έχουμε διάφορα για αυτή την κοινή συνεδρίαση. Όχι. <clears throat> Η ψηφοφορία θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου στις 9. Διάφορα όχι. Κλείνω την κοινή συνεδρίαση ΔΕΒΕ, ΕΝΒΙ και τα μέλη ένβη <clears throat> συγγνώμη, τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν. Αλλά ήσυχα παρακαλώ, διότι θα αρχίσει αμέσω ψηφοφορία.